Colleghi, colleghi, possiamo cominciare. Voglio informare la Commissione che il θα ήθελα να ανακοινώσω στην Επίτροπη ότι ο πρόεδρος Αλμπερτίνη, επειδή έχει υποχρεώσει στην Ιταλία, δεν μπορεί να παρευρεθεί, θα είναι μαζί μας το απόγευμα και θα ήθελα την συνεργασία σας έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στις εργασίες μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 17 και 15 μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης θα ψηφίσουμε για τους υποψηφίους για το βραβείο Ζαχάροφ και θα ήθελα να είσαστε παρόντες. Σε σχέση με τη διερμηνία υπάρχει σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες εκτός από τα δανέζικα και τα μαλτέζικα. Το άρθρο 147 θεωρεί, μάλλον δυνάμει του άρθρου 147, εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ε, διερμηνέων και μεταφραστών, τότε δεν μπορεί να υπάρξει διερμηνία σε αυτές τις γλώσσες. Ας ε, εγκρίνουμε τα πρακτικά της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 υπάρχουν αντιρρήσεις. Καμία αντίρρηση. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Δεν έχω να σας ανακοινώσω τίποτα ως προεδρεύων, ως ε, πρόεδρος. Τίποτα δεν έχουμε και στα διάφορα. Άρα εξετάζουμε τον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων θα πρέπει να έχουν, να διαθέτουν θεώρηση όταν περνάνε τα εξωτερικά σύνορα και τρίτες χώρες όπου οι πολίτες δεν έχουν αυτή την υποχρέωση. Θα είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία, γι' αυτό θα πρέπει να έχετε τη μαγνητική σας, την ηλεκτρονική σας κάρτα. Και σας υπενθυμίζω ότι η εισηγήτρια είναι η κυρία Σάρα Λάτφορντ, Και επί της ουσίας η κυρία Τάνια Φαζάν θα παρεμβεί επί της ουσίας. Εξετάσαμε το σχέδιο και τις ε, τροπολογίες και η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών ήταν η 1η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε μία σειρά τροπολογιών επί των οποίων πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια, στη Σάρα Λάντφορτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση στην Επιτροπή μας την προηγούμενη εβδομάδα όπου προσφέρθηκε όχι μόνο στεναρή υποστήριξη για το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε ε, σχετικά με την ελεύθερη ε, μεταβίβαση των ε, υπηκόων των Βαλκανίων βέβαια μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων κριτηρίων ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. Έτσι λοιπόν, βεβαίως και είχαμε μια συζήτηση επικοδομητική για την επίτευξη του στόχου. Κατά τα άλλα όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την άποψη εκείνη που ε, εγώ πιστεύω ότι δεν ε, ταυτίζεται με αυτά που είπε η κυρία Φάιν που και αυτή θα μιλήσει και είναι βασική συγγήτρια στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρώτα απ' όλα εμείς ε, πιστεύουμε ότι και οι πέντε χώρες ε, των ε, Δυτικών Βαλκανίων οι οποίες έχουν ενταχθεί στη διαδικασία σταθεροποίησης και καλύπτονται από τα συμπεράσματα της Θεσσαλονίκη, όλες αυτές θα πρέπει να επωφεληθούν από το να συμπεριληφθούν στο νομικό πλαίσιο που καλύπτει αυτός ο τροποποιημένος κανονισμός. Εγώ λοιπόν πιστεύω η άποψή μου για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η οποία παρουσιάζεται με την τροπολογία υπαριθμών 17 είναι η βασική τροπολογία έτσι ώστε να συμπεριληφθούν η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Αλβανία στο πλαίσιο αυτής της ε, τροπολογίας ε, σχετικά με τον κανονισμό. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής που θα αφορά στην εφαρμογή αυτής της άρσης θεώρησης για τις χώρες εκείνες που δεν θα έχουν καλύψει τα κριτήρια μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Αναφέρομαι βέβαια στην Βοσνία, Ριζεγοβίνη και στην Αλβανία. Αυτά όλα σημαίνουν ότι δεν είναι απαραίτητο την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα πρόταση από πλευρά Επιτροπή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε τώρα στο κοσυφοπαίδιο. Εδώ κλειδί είναι η τροπολογία μου υπαριθμών 7 και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος. Διάλογος για θέματα θεώρησης με το κοσυφοπαίδιο έτσι ώστε να υπάρξει και ένας ε, χάρτης πορείας για, τις, ε, για την απελευθέρωση σε διατάξεις φιλελεύθερη σχετικά με την ε, θεώρηση. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να επιδείξετε ως Επιτροπή κάποια ανοχή, κάποια κατανόηση. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν ανησυχίες από ε, για το πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια τέτοια διατύπωση η οποία θα έχει ως στόχο να είναι ρεαλιστική αφενός, αφετέρου όμως ε, θα αναγνωρίζει και τις ε, νομικές δυσκολίες όπως επίσης και, ε, και την άψη που φορά ε, στο ότι ε, πάρα πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του πεδίου. Θέλω λοιπόν να δείξετε κατανόηση. Αν δεν μπορείτε να με στηρίξετε στο να ψηφίσετε υπέρ της τροπολογίας υπαριθμών 7, Υπάρχει και η τροπολογία 8 βέβαια που είναι παρεμφερής, αλλά εν πάση περιπτώσει παρακαλώ πολύ όσοι θέλετε να με στηρίξετε να ψηφίσετε υπέρ τη 7. Κατά τα άλλα, μπορούμε να ρυθμίσουμε τι λεπτομέρειε στο πλαίσιο τη ε, Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, γιατί θα συνεχιστούν κάποιε συζητήσει, έτσι ώστε να καλυφθούν ε, όσο δυνατόν περισσότερο και να υπάρξει μια ρύθμιση για το 25 που να καλύπτει σχεδόν όλους γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πράγματι το 25 να ενταχθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Παρακαλώ λοιπόν κατανόηση επ' αυτού. Εξάλλου θέλω να σας πω ότι πρέπει επίσης ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να ρυθμίσουμε και την τελική διατύπωση που αφορά στους νομικούς όρους ε, σχετικά με την Βοσνία, Ζεγοβίνη και την Αλβανία. Όσοι συμμετέχετε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για το ε, πώς επάξουν τέτοιου νομικές ρυθμίσεις έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει φιλελευθερωποίηση στις αρχές του επόμενου έτους. Και πάλι σας παρακαλώ να με στηρίξετε. Να ε, ψηφίσετε υπέρ της 17 και βεβαίως ε, κατά τα άλλα μπορούμε να ρυθμίσουμε όλα τα υπόλοιπα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία ε, Λάτφορντ ως ε, εισηγήτρια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, πολύ στενή συνεργασία με την κυρία Σάρα Λάτφορτ και με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Νομίζω ότι η κυρία Λάτφορτ ε, κατέθεσε μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση για την ε, φιλελευθερωποίηση σχετικά με την θεώρηση. Και βέβαια θα ρυθμίσουμε πολλά θέματα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Εγώ ως εισηγήτρια για θέματα που έχουν σχέση με την θεώρηση αναφερθώ σε δύο θέματα, κυρίως όσον αφορά την νομοθετική έκθεση. Ε, Μακεδονία, Μαυροβούνη, Σερβία, 1η Ιανουαρίου 2010, έρεται η δέσμευση ε, της θεώρησης βίζα για την ε, Μακεδονία. Αυτά ήδη ε, κρίθηκαν γιατί πληρεί τι ε, προϋποθέσεις. Αυτό ήδη αποφασίστηκε και οι υπόλοιπε χώρες ε, σύντομα θα το πράξουν και αυτές και ελπίζω αυτό να το αναγνωρίσει η Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ε, σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Σαράγεβο την περασμένη εβδομάδα. Όπως ξέρετε, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Αλβανία δεν εγκρίθηκαν, δεν εξετάστηκαν από την Επιτροπή και τότε πράγματι δεν τα κριτήρια και σωστό ήταν αυτό. Όμως δυστυχώς υποτίμησαν τον κίνδυνο να ε, ριζώσουν περισσότερο οι εθνοτικές διαφορές στην περιοχή αυτή. Και θέλω να πω ότι η δύσκολη πολιτική κατάσταση θα επιδροθεί περαιτέρω αν τελικά δεν δοθεί τώρα ένα θετικό μήνυμα στις αρμόδιες αρχές, ε, γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πράγματι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Ο επικεφαλής της Επιτροπής της Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα πήγε στο Σαράγεβο και ε, συνεχάρει τις αρμόδιες αρχές ε, για την πρόοδο που έχουν σημειώσει. Πόρεσαν να καλύψουν το 90% των κριτηρίων σε λίγες μόνο εβδομάδες, άρα ο στόχος τους είναι σαφής. Όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Διαφθορά στο ξέπλυμα του χρήματος, στις δραστηριότητες των τρομοκρατών, συμφώνησαν ακόμα και στην ανταλλαγή ε, αστυνομικών στοιχείων. Δύσκολο το καθήκον, αλλά το συμμερίστηκαν όλοι. Πριν από μερικές εβδομάδες τα πράγματα έμειζαν διαφορετικά όταν η Κομισιόν ε, είπε, έδωσε το πράσινο φως ε, για μόνο τρεις χώρες και εξαίρεσε αυτές τότε θεωρήσαμε ότι η κατάσταση αυτή θα έφερνε τους Βόσνιους σε πολύ δύσκολη θέση και κατά κάποιον τρόπο θα τους ε, καθιστούσε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει λοιπόν να σας πω, αν δεν ε, επιταχυνθεί με συγχωρείτε η κατάσταση, αυτό θα πλήξει κυρίως τους νέους και τους φτωχούς. Την επόμενη εβδομάδα η Βοσνία Ερσεγοβίνη θα αρχίσει να εκδίδει τα βιομετρικά διαβατήρια. Δεν περιμένουν ότι θα υπάρξουν ε, προβλήματα. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν εκδώσει 65.000 διαβατήρια και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ε, μεταφέρουν ευχάριστες ειδήσει στους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα έχει φτάσει η στιγμή για να στελεί ένα νέο θετικό μήνυμα και ε, στην ε, δική μου την έκθεση το εκφράζω αυτό, το είπε και η κυρία Λάτσφορντ. Πρώτα απ' όλα προτείνω να τους προσφέρουμε μία δυνατότητα προσωρινά να τους μεταφέρουμε ήδη τώρα στο λευκό κατάλογο. Βεβαίω, οι διατάξει περί ε, βίζα, θεώρηση θα ισχύουν πλήρω όταν θα έχουν καλύψει όλα τα κριτήρια για τη θεώρηση. Ε, και τότε θα ξαναδούμε το όλο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ και στην ίδια την Επιτροπή να στείλει τους εμπειρογνώμονες στη Βοσνία Ερσεγοβίνη το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ήδη κατά τις αρχές του επόμενου έτους. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι και η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο, καλύπτει ήδη όλα τα κριτήρια όσον αφορά την ασφάλεια των διαβατηρίων. Έχει εκδώσει 150.000 ε, βιομετρικά διαβατήρια μόνο από τον Ιούλιο και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την λαθρομετανάστευση, την δημόσια τάξη και τα δικαιώματα των πολιτών. Θα ήθελα ε, να πω και μερικά λόγια για το Κωσυφοπαίδιο. Είναι το μόνο τμήμα των Δυτικών Βαλκανίων το οποίο εξαιρείται παντελώς από τη διαδικασία φιλελευθερωποίησης. Πολύ λεπτό το θέμα, το γνωρίζω και προσπαθούμε να βρούμε μια τέτοια λύση η οποία θα σέβεται τη θέση όλων των κρατών μελών. Και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε και μια λύση για τους ανθρώπους του κοσφοπεδίου. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για το πώς θα συμπεριλάβουμε το κοσφοπέδιο στη διαδικασία της ε, φιλελευθεροποίησης. Ίσως μπορώ να σας πω ότι τα Δυτικά Βαλκάνια, εγώ προσωπικά έρχομαι από τη Σλοβενία, είναι ένα μοσαϊκό. Είναι ε, μια σειρά από ψηφίδες όπου αν λείπει μια ψηφίδα διαταράσσεται η σφαιρικότερη εικόνα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σταθερότητας και πιο έντονη διαίρεση στην περιοχή. Για άλλη μια φορά λοιπόν θέλω να σας πω ότι μιλάμε για ένα βασικό δικαιώμα των ανθρώπων, το δικαίωμα του να ταξιδεύουν και όλα αυτά τα συνδέω και με μια επιστολή που πήρα από έναν φοιτητή από τον Μπίχατς που είναι κοντά στη Σλοβενία, ο οποίος μου έγραψε ότι η Σλοβενία λόγω των ε, ε, συνόρων ε, του μοιάζει να είναι πολύ μακριά και λέει ότι η νέα γενιά στις όμορες χώρες θα ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνοι μπορούν να ταξιδεύουν ενώ οι ίδιοι είναι ε, όμοιροι της πολιτικής. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή όπου να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους πολίτες του Ανατολικού Βαλκανίων ότι όλοι πλέον έχουν το ίδιο δικαίωμα, δηλαδή να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έναν κατάλογο, μεγάλο κατάλογο συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Θα ήθελα να περιοριστείτε στο χρόνο ομιλία σας, έτσι ώστε να επιτρέψουμε σε όλους να εκφραστούν. Η κυρία Πακ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να πω το εξής. Το ζήτημα της ελευθέρωσης της θεώρησης δεν έχει καμία σχέση με τη συζήτηση για τη διεύρυνση. Παρακαλώ να το σκεφτείτε. Όταν υπήρχε η Ιουκοσλαβία ακόμα, όλοι οι Ιουκοσλαβοί μπορούσαν να ταξιδεύουν. Δεν είχαν το πρόβλημα που έχουν σήμερα. Κανένας από αυτούς. Παρακαλώ προσπαθήστε να κάνετε μία ε, διάκριση ανάμεσα στην οριμότητά τους να μπουν στην Ευρώπη και στην οριμότητά τους να βγουν από τη θεώρηση διαβατηρίων. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και συμφωνώ και με την προλαλή σας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ε, στη μεταχείριση από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αν η Σερβία και το Μαυροβούνι δεν πληρούν ακόμα τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να έχουν την ίδια μοίρα με κάποιους άλλους, δηλαδή στο ίδιο πλαίσιο. Σερβία και Μαυροβούνι θα πρέπει ταυτόχρονα να λέμε και Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη και αυτές δεν τηρούν ακόμα όλες τις προϋποθέσεις αλλά από τον Ιούνιο και στις δύο αυτές χώρες έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Υπογραμμίζω όλα αυτά που υπόθηκαν για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, τα είπα ήδη την προηγούμενη φορά. Ωστόσο επιτρέψτε μου να πω ότι ξεχνάμε πάντα ότι η Αλβανία είναι μια χώρα πάρα πολύ σταθερή, με σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό μετά τις τελευταίες εκλογές που ποντάρει πάρα πολύ για να γίνει και όριμη να μπει στην Ευρώπη. Πάνω από 150.000 βιομετρικά διαβατήρια έχουν εκδώσει από τον Ιούνιο. Ε, Κάποιε άλλε χώρε ακόμα δεν το έχουν κάνει αυτό. Παρακαλώ θερμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κάνει εδώ διακρίσει. Διότι έτσι αντιβαίνει και αντιφάσχει με την καλή βούληση και πίστη και ε, αυτό που μπορεί κανείς να περιμένει από εμάς στην Ευρώπη. Αλβανία και Βοσνία, Ζεγοβίνη τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ίδια μεταχείριση με τα υπόλοιπα τρία κράτη και το επέδειο λόγω της ιδιαιτερότητάς τους με τις τροπολογίες μας πιστεύω το έχουμε καλύψει. Τις υποστηρίζω πλήρως και Κάπω ε, σωστά έχουμε τακτοποιήσει και αυτή την περίπτωση. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε εκεί μαύρη τρύπα για ε, την ε, απαλλαγή θεώρηση. Και επίσης θεωρώ, σε αντίθεση με την τροπολογία 18 δυστυχώ που τα γράφει αυτά, δεν θα πρέπει να καλέσουμε και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Χρόνου να ξεκινήσει και πάλι νομική διαδικασία. Όχι! Τώρα θα πρέπει να υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν για τη ε, Βοσνία Ζεγοβίνη, για τη Σερβία το Μαυροβούνιο και να πούμε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μπορούν να ε, ενταχθούν τότε και τότε και όλα αυτά να ελεγχθούν χωρίς να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία. Αυτό θα σημαίνει τεράστια αλληγόρια. Ε, γι' αυτό διαφωνώ με την τροπολογία 18 και ελπίζω να περάσει η 17. Αυτά, Πρόεδρε, τα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε μια νέα συζήτηση επί του θέματος και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, διότι όλοι μας είμαστε πολύ απασχολημένοι σήμερα. Αλλά ως συντονητής των σοσιαλιστών και δημοκρατών και ως κοιόδης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βαρόνι Λάτφορτ, διότι συνεργάστηκε με τη ΛΥΜΠΕ. Η συνεργασία αυτή είναι ύψη της σημασίας έτσι ώστε να στείλουμε τα σωστά μηνύματα με βάση την έκθεση της ΛΥΜΠΕ και της ΑΦΕΤ συμβαδίζουμε με την, κυρία Λάτφορντ και την κυρία Φαγιόν. Θεωρούμε ότι όλες τις χώρες θα πρέπει να τις εντάξουμε στη νομοθετική διαδικασία όπως ορίζει η Επιτροπή, δεν θα ήθελα να επαναλάβω όσα προελέχθησαν. Ως προς το κοσυφοπέδιο, θα θέλαμε να υπάρχει μία λίγο τροποποιημένη θέση Δεν είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την τροπολογία της ε, κυρίας Λάτφορ, την 7 δηλαδή. Θα θέλαμε να υποστηρίξετε την 5 που αποτελεί ένα συμβιβασμό που μπορεί να υποστηρίξει η ΑΦΕΤ στο σύνολό της. Ορισμένοι συνάδελφοι υπέβαλαν άλλε τροπολογίε με ελεύθερη ψηφοφορία, με ελεύθερη ψήφο, αλλά νομίζω ότι αυτή η τροπολογία μπορεί να υποστηριχθεί από όλου. Τέλος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Αλβανία, ε, ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Βοσνία μετά την πρόταση της Κομισιόν και πρέπει να υποστηρίξουμε την περιφέρεια, διότι το θέμα της ελευθέρωσης των θεωρήσεων είναι, αποτελεί το επίκεντρο της, ε, των, της έγνοιας των πολιτών, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών και άρα θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Πρόεδρος, όταν δίνω το λόγο δεν ξέρω ποιο θα είναι το περιεχόμενο της παρέμβασής τους. Δεν θα ήθελα να ανοίξω συζήτηση και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όσους ε, ζήτησαν να παρέμβουν να παραμείνουν στην ουσία του θέματος, δηλαδή την ε, ψηφοφορία επί των τροπολογιών και να μην ε, ξανανοίξουμε μια συζήτηση που έχει προηγηθεί. Ευχαριστώ. Τάλερ. Θα είμαι πολύ σύντομος, ιδιαίτερα γιατί κατανοώ ότι θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε αμέσως ως ε, πολίτης της πρώην Ιουκοσλαβίας μπορώ να σας πω ότι 20 χρόνια πριν η κατάσταση ήταν πολύ εύκολη για μας. Δηλαδή μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στην Τεργέστη, στη Βενετία, στη Θεσσαλονίκη, στο Γκράτς 25 χρόνια δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στη Σόφια, Βουδαπέστη και Βουκουρέστη, δηλαδή στην πρώην δημοκρατία της Ιουκοσλαβίας. Μπορούσαμε, είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε στη Δύση ελεύθερα. Τώρα λοιπόν επανερχόμαστε σε αυτή την κατάσταση έτσι ώστε η νέα γενιά να νιώσει πώς ήταν η κατάσταση 25 χρόνια πριν. Ας υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Αποστέλουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα στην περιφέρεια που είναι πολύ μεγάλη σημασία ως προς το κοσυφοπαίδιο. Η πρότασή μου είναι η εξής. Ας ξεχάσουμε το νομικό υπόβαθρο που αφορά το κοσυφοπαίδιο. Εμείς το κάνουμε αυτό για τους ανθρώπους που ε, ζουν εκεί. Πρόκειται για πολίτες που έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αναγνωρίζεται το κοσυποπέδιο από όλα τα κράτη-μέλη. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επί της ουσίας των τροπολογιών. Να σχολιάσετε μόνο τις τροπολογίες σας, παρακαλώ. Van Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω και εκτιμώ τη δουλειά της συναδέλφου μου Σάρα Θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν στέλνουμε απλώ μηνύματα στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά στέλνουμε μηνύματα και στου λαού των 27 κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούμε να καταπολεμούμε ε, τη λαθρομετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Μπορεί να μου εγγυηθεί η εισηγήτρια ότι δεν πρόκειται καμία χώρα να έχει τέτοιο καθεστώς απαλλαγής ε, από τη θεώρηση αν δεν πληρεί όλα τα κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Μποσκούρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η γραμμή που ακολούθησε η συγγήτρια κυρία Λάτφορτ και ε, ε, της ουσίας ε, φαγιών στη Λίβε είναι πολύ καλή, λογική. Θα πρέπει να μην κάνουμε διακρίσεις μεταξύ Σέρβων, Κροατών και Βοσνίων, να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και ισότιμη, βεβαίως τα κριτήρια, αλλά να μην τους αποκλείουμε από χέρι. Και όλοι στο Κοινοβούλιο μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή και διοικητικό φόρτο. Εφόσον πληρώνουν λοιπόν τα κριτήρια, θα πρέπει οι χώρε αυτέ να βγουν από το καθεστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κάτσιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μας υπενθυμίσω σε όλους μας το ρόλο του Κοινοβουλίου. Εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε τον δυναμισμό, αυτό τη δυναμική πορεία στην περιφέρεια. Η ΑΦΕΤ και η ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτούς τους προκριματικούς όρους, ας το πω έτσι, για να υπάρχει αυτός ο δυναμισμός σε μεμονωμένες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις στην περιφέρεια που τίθενται υπέρ της Ευρώπης. Το θέμα της ε, ε, Βοσνίας Ερζεγοφίνης είναι το πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα μπορεί όμως να επιτελέσει πρόοδος βραχυπρόθεσμα, δηλαδή άμεσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το, τις συναδέλφους Φαγιών και Λάντφορτ για την εργασία τους και θα ήθελα να τονίσω ότι οι μηνιαίες αξιολογήσεις της Επιτροπής, δηλαδή τροπολογία 2 εδάφιο 4, είναι ύψης της σημασίας. Η Αλβανία θα ακολουθήσει άμεσα. Αλλά κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι το κοσυφοπαίδιο δεν μπορούμε πλέον να το αγνοήσουμε. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο και τους πολίτες του, όχι ως χώρα, αλλά θα πρέπει να μας ε, απασχολούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών από το κοσυφοπέδιο. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε πλέον. Δεν μπορούμε να βάζουμε κατά μέρο τα συμφέροντα αυτών των πολιτών. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να είσαστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ζητώ την κατανόησή σας. Λένερ. Μαντλένερ, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος κι εγώ. Ακούω πολλά που λένε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ε, είναι κάτι το οποίο παραβιάζεται από τη θεώρηση διαβατηρίων. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ποιο ζητάει βίζα την παίρνει. Μην θεωρούμε ότι είναι κλειστά τα σύνορα. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι μπορούν να ε, ταξιδεύουν. Μόνο οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες πλήττονται και είναι λάθο το μήνυμα, ενθαρρύνουμε του τρομοκράτε και τους εγκληματίες αν καταργήσουμε τη βίζα προς τις χώρε αυτές. Ο κανονικός κόσμος, οι φυσιολογικοί άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν θεώρηση και να την πάρουν. Για διαδικαστικό. Ο κύριος έχει το λόγο για διαδικαστικό. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την μερίσια διάταξη που εγκρίναμε στην αρχή της συνεδρίασης, βλέπω ότι δεν προβλέπεται συζήτηση για την έκθεση και τώρα γίνεται συζήτηση. Συζήτηση επί της έκθεσης. Εάν γίνει και εφόσον θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρευρισκόμαστε στην αίθουσα για τη διενέργεια της ε, ψηφοφορίας και μόνο γι' αυτό και θα πρέπει να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα, να το ψηφίσουμε, να μην το συζητήσουμε. Διαφορετικά αλλάξτε την ημερήσια διάταξη, εάν, αν πρόκειται να γίνει συζήτηση. come... Όπως ήδη είπα, είναι πολύ δύσκολο να λογοκρίνω τους συναδέλφους γιατί θεωρητικά οι συνάδελφοι θα πρέπει να μιλήσουν επί της ουσίας των τροπολογιών εντάχει. Εάν όμως ε, συμφωνεί ολόκληρη η Επιτροπή, ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ του να προβούμε στην ψηφοφορία άμεσα. Να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Η συγγήτρια ζήτησε το λόγο. Η κυρία Λάντφορτ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, θα ήθελα απλά να πω, να απευθυνθώ στο συνάδελφό μου Βαν Πάολεν και να δώσω και μία απάντηση σε αυτά που είπε ε, τον κύριο Ματλένα ότι ε, αν όμως εξαιρεθούν κάποιοι από την θεώρηση αυτό ευνοεί τους τρομοκράτες. Κοιτάξτε, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να άρουμε την υποχρέωση θεώρησης ε, εάν δεν καλύπτονται τα κριτήρια για τη λαθρομετανάστευση, για τις προϋποθέσεις εισδοχής σε μια χώρα, για την δικαστική συνεργασία, και για την συνεργασία κρατών για την επιβολή του δικαίου. Μόνο έτσι κανεί μπορεί να αντιμετωπίσει του ε, τρομοκράτε. Και αυτό κάναμε στο ΕΒ όταν είχαμε την ε, ελεύθερη μετακίνηση με του Ιρλανδούς. Ε, ποτέ δεν σταμάτησε η ελεύθερη μετακίνηση γιατί απλά υπήρχε συνεργασία ανάμεσα σε αστυνομικέ αρχέ που οδηγούσε στη σύλληψη των τρομοκρατών. Με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει το θέμα. Επουδενή όμω δεν πρέπει να αμβληνθούν τα κριτήρια γιατί αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για μας αλλά ούτε και για τους ίδιους. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Εάν η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θεωρεί ότι θα έπρεπε άμεσα να προβούμε στην ψηφοφορία, να σηκώσετε το χέρι. Ποιοι είναι υπέρ της άμεσης ψηφοφορίας. Νομίζω ότι καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία. Άρα δεν σας δίνω πλέον το λόγο και δεν σημαίνει ότι δεν είμαι αυρός κάνοντάς το. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 17, τροπολογία 17 τη συναδέλφου Λάντφορτ. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ της 17 παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 18. 19 μάλλον, Λάντφορτ. 19, υπέρ της 19 παρακαλώ. 19, 19, 19, 19. Όχι 18, 19. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. L'emendamento eh, Τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Επαλήθευση λοιπόν με ηλεκτρονική. Παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά επί της 4. Υπάρχουν προβλήματα. Abstention. Εσείς τι ψηφίζετε, αποχή. Αποχή ή αρνητική ψήφος. Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος που έχει πρόβλημα με την ηλεκτρονική του κάρτα. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συνάδελφος εκφράστηκε αρνητικά δεν έχει πρόβλημα με την κάρτα της. 7. Λάντφορντ. Θα ήθελα να ψηφίσετε τώρα ποιοι τάσσονται υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ωραία, ψηφίστε. Ψηφίζουμε τώρα. Chiudiamo il Πέρας. È adottato. Εγκρίνεται. Quindi possiamo... Allora si aggiunge un voto favorevole. Προσθέτουμε μια θετική ψήφο. You in favor? Είστε υπέρ, εντάξει. Με συγχωρείτε, με Έχουμε άλλη μία ψήφο υπέρ και μία κατά. Δεν μπορεί να... Ε, ψήφισε κατά ο συνάδελφος ε, διότι δεν ε, λειτουργεί η κάρτα του. Ωραία. Άρα εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι, Κύριε Πρόεδρε, ε, Νομίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Βρισκόμαστε στην 6, τροπολογία 6. Υπέρ. 6. 6. Chi è a favore? Κατά. Ωραία, ηλεκτρονική. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε ηλεκτρονικά επί της 6. Πέρας. Έχω τώρα την ε, ηλεκτρονική μου κάρτα, αλλά του συναδέλφου δεν ε, λειτουργεί και τάσεται υπέρ. Ναι, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Εντάξει, καταγράφουμε την ψήφο του συναδέλφου, αλλά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. 9 με μια προφορική. Ποιοι τάσσονται υπέρ της 9 κατά εγκρίνεται. Τώρα οι δύο. Ποιοι τάσσονται υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Ε, δεν έχει σημασία γιατί απορρίπτεται κυρία Πακ. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ας επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ποιοι τάσσονται υπέρ. Και Κατά. Πρέπει πάντα, α, μάλλον συγγνώμη, ψηφίζουμε με ηλεκτρονική, έκανα εγώ λάθο, λέει ο πρόεδρο. κλείνουμε την ψηφοφορία. Ερεσπίντο. Siamo al 15. Απορρίφθηκε. 15. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ τη 15, κατά. Απορρίπτεται. Τέλος, τροπολογία 16. Παρακαλώ, ποιοι τάσσονται υπέρ, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Α, η κυρία Λάτφορντ. Έχετε το λόγο, κυρία Λάτφορντ. Κοιτάξτε, απλά θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, όπως είπα και πριν από την ψηφοφορία ότι το θέμα του κοσμοπεδίου είναι πολύ ευαίσθητο και θα ήθελα ε, να δείξετε κάποια κατανόηση. Ε, βεβαίως ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει δίσταντη απόψη για την 5 ήταν τσίμα τσίμα ε, το αποτέλεσμα της ψηφορίας. Θα ήθελα λοιπόν να μην επηρεάσετε απαραίτητα όσοι διαφωνείτε το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί βρίσκεται στα χέρια της κυρίας Φάιλε και τελικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα λεπτά θέματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσπαθήσετε να έχετε αυτά κατά νου που σας είπα. Να ξέρετε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων στην Επιτροπή. Ε, περίπου με απόλυτη ισορροπία. Επειδή εγώ όμω ε, είμαι και στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, ό,τι διαφωνία υπάρχει εδώ θα προσπαθήσουμε εκεί να το ρυθμίσουμε. Τελική ψηφοφορία. Πάντα ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Chiudiamo la votazione. Eras. Il provvedimento adottato Ωραία, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. E και να συγχαρούμε και την κυρία Λάτφορντ. Και το σκάμπιο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 να διαμαρτυρηθώ για το πώς διαχειριστήκατε πριν τις παρεμβάσεις, διότι επιτρέψατε να παρεύουν τα μέλη της Επιτροπής, ένα μεγάλο μέρος, εκτός από αυτούς που παρέμεναν. Δηλαδή, είτε γίνεται συζήτηση, είτε δεν γίνεται, δεν μπορείτε να την αφήνετε στη μέση, διότι έγινε διάκριση κατά των μελών που δεν εκφράστηκαν. Και θα ήθελα να, να εκφράσω τη διαμαρτυρία μου για το πώς διαχειριστήκατε το θέμα. Υπήρχαν διαφορετικές ε, τροπολογίες από την ε, πλειοψηφία και θα ήθελα να εκφραστώ για δύο τροπολογίες που δεν πρόκειται για, μάλλον σε σχέση με το κοσυφοπέδιο δεν μιλάμε για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους Κωσοβάρους. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές για να διαχειριστούν και να διαπραγματευτούν αυτές τις ε, θεωρήσεις δεν, έχει, ε, δεν σχετίζεται με τους Κωσοβάρους, αλλά με το ποιοι είναι υπεύθυνοι με τους οποίους πρέπει να διαπραγματευτούμε αυτές ε, τις θεωρήσεις. Δηλαδή, έχουμε την, το ψήφισμα 1245 για το ποιες θεωρούνται οι αρμόδιες ε, αρχές διαπραγμάτευσης του καθεστώτος του Κωσυφοπεδίου και αυτό δυνάμει του ψηφίσματος 1245 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συνάδελφοι. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση, αλλά μπάση περιπτώσει ε, αρκέστηκα στην πλειοψηφία. Ναι, εντάξει. Δεν μπορείτε να σταματήσετε όμως τη συζήτηση στη μέση, δηλαδή όταν μίλησαν μόνο αυτοί που τάχθηκαν υπέρ ορισμένων θέσεων. Ωραία, τι να κάνω, λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις σας και θεωρώ ότι πράγματι αυτό έγινε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Έκβαση του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο πρόεδρος Αλμπερτίνη έκρινε σκόπιμο να το εγγράψει στην ημερήσια διάταξη. Πριν εξετάσουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κοινή Δράσης που αφορά τον συνάδελφο Νέτς. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Εδώ εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις για την ε, παρούσα κατάσταση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και για το μέλλον τους. Είμαστε όμως όλοι ενωμένοι θεωρώντας ότι οι δημοκρατικές αρχές ε, υπερέχουν και βεβαίως και η λαϊκή βούληση. Άρα με βάση αυτή την αρχή θα εργαστούμε για την καλύτερη διεκπαιρέωση των θεσμικών μας ε, ζητημάτων. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας κύρωσης της συνθήκης όπου θα πρέπει να βρούμε ευέλικτες και πραγματιστικές λύσεις σε σχέση με τις καθυστερήσεις που επήλθαν για την κύρωση της συνθήκης. Νομίζω ότι γνωρίζετε το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τσεχίας, ο κύριος Κλάους, δεν έχει εκφράσει τις προθέσεις του για το πότε θα γίνει η κύρωση, όπως ορίζουν ορίζει και η Γερουσία και η Βουλή της Τσεχίας, διότι όπως ξέρετε έχει γίνει μια προσφύγη στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας από ορισμένους γερουσιαστές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσει κατά μερικές εβδομάδες ή μήνες η ισχύ της συνθήκης. Άρα, εν ώψη της συζήτησης που θα γίνει στην Ολομέλεια, αυτή τη βδομάδα θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας ως ΑΦΕΤ. Σας προτείνω λοιπόν ορισμένα ζητήματα και θα δώσω το λόγο στους συντονιστές ή στους εκπροσώπους τους για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Καταρχήν, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ε, ε, λειτουργησιμότητα των θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, θεσμικές ε, καινοτομίες, διότι η συνθήκη της Νίκαιας προβλέπει μείωση του αριθμού επιτρόπων 26 και όχι 27, ενώ η συνθήκη της Λισαβόνας ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να ισχύει ένας επίτροπος ανακράτος μέλος, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μερικοί πιστεύουν ότι η λύση θα ήταν να διοριστεί η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος με την θέση σε ισχύ χωρίς να λάβουμε υπόψη το πότε θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και από το αποκλεισμένο κράτος μέλος του Διευθυντηρίου θα δώσουμε το, το λειτουργήμα, την, τη θέση του ύπατου. Εάν ε, ισχύσει κάτι τέτοιο, το ζήτημα είναι τι θα γίνει τη στιγμή της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Τι θα γίνει τότε η ε, ε, παρέτηση του, του Επιτρόπου Ρέλεξ θα σχετίζεται με έναν ανασχηματισμό των ε, χαρτοφυλακίων και οι αρμοδιότητες των επιτρόπων ορίζονται ανάλογα με τα χαρτοφυλάκια. Ένας ανασχηματισμός λοιπόν ε, ίσως οδηγεί σε ψήφο εμπιστοσύνης. Άλλο θέμα. Πώς θα διοριστεί ο ύπατος εκπρόσωπος θα δεχόταν την αρχή του να ε, γίνει ακρόαση ενώπιον του Κοινοβουλίου πριν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτά τα σημεία και δίνω το λόγο σε όσους θα ήθελα να παρέμβουν και θα σας ακούσω όλους με μεγάλη προσοχή. Νέτς. Κυρία Νέτς, ευχαριστώ. Thank uh, Στα αγγλικά η κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα εξ ονόματος των συναδέλφων της πολιτικής μου ομάδας να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση για την έκβαση του δημοψηφίσματος στην Ελλαδία. Ε, πάνω από 67% ε, ψήφισαν υπέρ της σύνθηξης της Λισαβόνας και αυτό είναι πραγματικά νίκη για την Ευρώπη. Εδώ είναι και παράδοξο το γεγονός ότι ο Ιρλανδικός λαός κατάλαβε πλήρως τι σημαίνει το να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περνώντας όλα τα δεινά και τα βάσανα από τη βαθιά οικονομική κρίση. Αυτό φαίνεται ήταν το αποφασιστικό ε, που τους έκανε να αλλάξουν γνώμη και να υποστηρίξουν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη και δεν μπορώ παρά να Ελπίζω ότι οι δύο πρόεδροι των κρατών μελών που ακόμα δεν έχουν κυρώσει ε, τη συνθήκη που έχει ε, κατά τα άλλα περάσει τη διαδικασία κύρωση σωστά από τα κοινοβούλια του. Ελπίζω να υπογράψουν και οι δύο πρόεδροι για να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη. Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα καλά. Ε, θέλετε από μένα τώρα να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ή να περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμα, να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλετε να μιλήσω εγώ και να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου. Όχι, για τη Λισαβόνα λοιπόν. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή στεθεί σε ισχύ θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Από τις σημαντικότερες βεβαίως είναι ότι θα υπάρχει εξαφάνιση της διάκρισης μεταξύ των τριών πυλώνων, πολύ ε, σημαντικό. Θα έχουμε πολύ περισσότερη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία, αλλά και ε, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας θα επέλθουν οι μεγαλύτερες αλλαγές. Με τη δημιουργία Μάλλον να το πω αλλιώς. Ε, πρώτον, τις θέσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα εκπροσωπεί προς τα έξω σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη θέση του ε, υπάτου εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που ταυτόχρονα θα είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα που θα το βρούμε αυτό το καταπληκτικό ή την καταπληκτική προσωπικότητα είναι άλλη υπόθεση. Αλλά υπάρχει μια σύνθεση. Ο ύπατος εκπρόσωπος εργάζεται σε πολύ στενή συνεργασία με το Συμβούλιο από τη μια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη, εφόσον και αντιπρόεδρός της. Uh, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και θα επιτρέψει πραγματικά να γεφυρωθεί ένα χάσμα που καμιά φορά στο παρελθόν υπήρχε. Και τέλος δημιουργείται μια υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εμβαθύνω σε λίγα λεπτά θετικά Και αυτή τη στιγμή θέλω να ε, χρησιμοποιήσω μια ουδέτερη έκφραση, η ανάπτυξη, για να το χαρακτηρίσω έτσι, ε, μια διπλωματική υπηρεσία και διπλωματική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι από τι μεγάλε προκλήσει για τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπρόκ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω και εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα με 67,1% είναι εντυπωσιακό όχι μόνο για την Ιρλανδία αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποδεικνύεται ότι μέσα από μία μακρά συζήτηση αν μπορεί κανείς ε, να εξηγήσει τα πράγματα ε, όπως ακριβώς αναφέρονται στη συνθήκη, τότε οι πολίτες ε, τα δέχονται και με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε αυτές τις αιτιάσεις που εκτοξεύανταν ε, λόγω της κακής ε, ερμηνείας συνθήκης να αποδείξουμε ότι όλα αυτά δεν υφίστανται, δεν έχουν καμία σχέση με την συνθήκη. Κατόπιν τούτου πρόκειψε μια νέα συζήτηση στην Ιρλανδία όπου οι αγωνίες των Ιρλανδών ελήφθησαν υπόψη χωρίς να τροποποιηθεί η συνθήκη. Γιατί δεν ήταν απαραίτητο κάτι τέτοιο. Απλά δόθηκαν απαντήσεις ε, στις ε, στην κατασυκοφάντηση της ε, συνθήκης. Αυτή τη φορά, εν πάση περιπτώσει, η συνθήκη ενεκρίθη και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μία ένδειξη για το ότι η ε, διαδικασία επικύρωσης μπορεί να συνεχιστεί με επιτυχία. Και βλέπουμε ότι από την ε, Παρασκευή η συνθήκη σε όλες τις χώρες έχει επικυρωθεί πλέον ε, είτε με κοινοβουλευτική διαδικασία είτε με οποιαδήποτε άλλη. Και λείπουν οι υπογραφές έξι μη εκτελεστικών πρόεδρων. Αυτό έχει σημασία για τη συνθήκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούμε από την Πολωνία ότι ο κ. Κασίνσκι, ο Πολωνός Πρωθυπουργός, ε, άφησε να εννοηθεί ότι θα τηρήσει το λόγο του και μετά το Ιρλανδικό δημοψήφισμα ε, θα υπογράψει. Έτσι και λέω, εγώ δεν περίμενα τίποτα άλλο και νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή επισήμανση έτσι ώστε η συζήτηση παραμένει απαραίτητη μόνο σε μία και μόνο περίπτωση. Και θεωρώ ότι όλα αυτά ε, πρέπει να τα κάνουμε με την ησυχία μας, να περιμένουμε την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, να δούμε τι θα κάνουμε. Πράγματι η συνθήκη πρέπει να συμβαδίζει ε, με, την, ε, με το Σύνταγμα της Τσεχίας. Δεν νομίζω ότι εκεί θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα και ως εκ τούτου ε, θεωρώ ότι επειδή δεν θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ, σύντομα θα, θα μπορούμε να έχουμε και την υπογραφή έτσι ώστε μέχρι το τέλος του έτους η συνθήκη να μπορεί να τεθεί σε ισχύ. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, το οποίο με απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Υποτίθεται υπάρχει μια επιστολή ε, της αντιπολίτευσης μιας χώρας που έχει ήδη επικυρώσει τη συνθήκη και μάλιστα ε, με δοσμοφτικό χαρακτήρα, ο οποίος λέει στον πρόεδρο μιας άλλης χώρας να μην ακολουθήσει την πρόταση του Κοινοβουλίου και του δικού του του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ε, πώς μπορεί κανείς να αντιδράσει στην επιστολή ενός τέτοιου αρχηγού αντιπολίτευσης, αν ας πούμε ο αρχηγός αντιπολίτευσης στη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Ολλανδία στέλνει μια επιστολή ε, ας πούμε στη Βασίλισσα της Αγγλίας, παρακαλώ μην υπογράψετε τον νόμο ή την πρόταση που σας στέλνει η Βουλή. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και μπορώ να φανταστώ πώς θα αντιδράσει ο Βρετανικός τύπος, όπως τον γνωρίζουμε. Και νομίζω λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει στη συζήτησή μας, χωρίς βέβαια να ε, εκνευριστούμε, γιατί εδώ πρόκειται για θέση του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν θα αποτελέσει κριτήριο για την απόφαση του Πρόεδρου ε, Κλάους. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί ο Πρόεδρος από αυτήν την ε, επιστολή και θεωρώ ότι τελικά θα δώσει την υπογραφή του. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έχουν σχέση ε, με το Σύνταγμα, αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγει με βάση τη συνθήκη της Νίκαιας και λόγω των ημερομηνιών που υφίστανται Ίσως ε, θα πρέπει να αφήσουμε να τρέξει η κανονική διαδικασία και ε, όπως ε, σας είπα μπορούμε το χρονοδιάγραμμα να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος του έτους για να καλυφθούν οι θέσεις της Κομισιόν, έστω και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και κατόπιν, όσον αφορά τον ύπατο εκπρόσωπο, να προσθεθεί μια διαδικασία με την έννοια ότι ε, θα πρόκειται για τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Με βάση τις απόψεις του Κοινοβουλίου, ο ύπατος εκπρόσωπος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως οποιοδήποτε άλλος επίτροπος. Για να φτάσει εκεί είναι πολύ πιο μακρύς ο δρόμος. Ε, χρειάζεται την απόφαση του Συμβουλίου, ε, χρειάζεται και πολλές άλλες διαδικασίες, αλλά εν πάση περιπτώσει όσον αφορά την αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο. Ε, το Κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά, του είναι παντελώς αδιάφορο. Και επ' ε, και με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε, να δούμε τι σημασία έχουν όλα αυτά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να τηρήσουμε ή να εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να μην παραδώσουμε εδώ ένα ατού το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ. ο συνάδελφο Μέγερ, γιατί είπατε ή συνάδελφο Μέγερ, πρόεδρε. Πρώτον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για δεύτερη φορά καλείται να ψηφίσει ο λαός της Ιρλανδίας. Την πρώτη φορά ψήφισε όχι. Ε, τώρα ψήφισε ναι βέβαια. Ε, και είναι γεγονός και θα ήθελα να σας θέσω υπόψη το εξή. Αν είχε βγει το όχι, θα κάναν και τρίτο και τέταρτο μέχρι να βγει το ναι. Περίεργοι κανόνες παιχνιδιού είναι αυτοί που βάλαμε στο τόσο περίπλοκο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την εκφράζω αυτή την κριτική εξ ονόματος μιας ε, ε, κοινοβουλευτική ομάδας που δεν είναι ευρωσκεπτικιστική, είναι ευρωαπαιτητική. Και για να έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα, θα πρέπει να είναι πλήρη ο σεβασμός τη δημοκρατία και των πολιτών. Και τι δείχνει αυτό. Και στην περίπτωση αυτή, όπω είδαμε, ο Ιρλανδικός λαός υπέστη μια δεύτερη προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ιρλανδικές εταιρείε έχουν ξοδέψει τεράστια ποσά και ήταν τελείως άνηση η όρη της προεκλογικής εκστρατείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τι δείχνει, ότι μέχρι ποιο βαθμό αυτό το οικοδόμημα χωλαίνει και πάει σε μια κατεύθυνση τελείως στραβή. Αν θέλουμε πραγματικά να ε, οικοδομήσουμε ένα κοινό χώρο που μας ενδιαφέρει να συμμετέχουν οι πολίτες και όλο περισσότεροι να είναι η ε, Ευρώπη συνεκτική, κοινωνική και ίση. Έτσι λοιπόν, ούτε η στρατηγική της Λισαβόνας που ισχύει, που υποτίθεται ότι θα έφτανε στο 3% ε, και η ανάπτυξη ε, με 20 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και στην καινοτομία και στην έρευνα να επενδύεται το 3%. Λοιπόν, η περίφημη αυτή η στρατηγική της Λισαβόνας όχι μόνο δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στη χειρότερη κατάσταση που γνώρισε η Ευρώπη από το 30 στην οικονομική δραστηριότητα και ε, στους δείκτες απασχόλησης. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Αν αυτή η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε, γιατί κανένας δεν αναβάνει την ευθύνη. Ερώτηση δεύτερη. Αφού φτάσαμε εδώ, και έχουμε τη συνθήκη της Αβώνας που ε, προωθεί ένα οικονομικό μοντέλο ε, το οποίο ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, βλέπε άρθρα 43 έως και 49 που στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έτσι, δικαιολογούν αποφάσεις για το κοινωνικό dumping, κοινωνικό dumping στην Ευρώπη που καταστρέφει όλες τις κοινωνικές αξίες. Και παρόλα αυτά τα δύο άρθρα αυτά, το 43 και το 49, βάζουν τα θεμέλια για τη Λισαβόνα και ε, λένε ότι η άκρητη λειτουργία της αγοράς, η άκρατη και αχαλήνοτη λειτουργία της αγοράς επικυριαρχεί των δικαιωμάτων των πολιτών και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Και η δική μας πολιτική ομάδα ρώτησε τον κύριο Ντουράου Μπαρόσο πριν εκλεγεί γιατί δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτυχίας της στρατηγικής Λισαβόνας και μας απάντησε ε, με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν αναβάνω την ευθύνη διότι φταίει η οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λες και εδώ η συνένεση της Ουάσιγκτον δεν είχε εφαρμοστεί ε, τα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν με την αγορά να την αφήσουν ε, ελεύθερη. Μα η μέθοδος για να χτιστεί η Ευρώπη και το περιεχόμενο των συνθήκων απέχουν όλο και περισσότερο από την ανάγκη να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και πιο κοινωνική Ευρώπη. Για να μην έρθω και στην εξωτερική πολιτική. Και θέλω εδώ να επικρίνω λίγο τη γραμματεία. Δεν επιτρέπεται χτε να μα έρχεται ένα έγγραφο για την εξωτερική υπηρεσία για να ψηφίσουμε αύριο. Μάλλον να λύγει η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών την επομένη. Αυτό είναι τελείω απαράδεκτο. Και μιλάμε και για τέτοια έκθεση της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείτε να μας δίνετε τη μια μέρα το κείμενο και την άλλη μέρα να έχουμε κάνει τις τροπολογίες μας. Ε, κατηγορηματικά καταγγέλνουμε αυτή τη μέθοδο. Δεν είναι μέθοδοι αυτές και ε, περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι τροπολογίες γιατί μιλάμε για κάτι σημαντικό. Και για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην καταρτίζεται ημερήσια διάταξη από τις Ηνωμένε Πολιτείες ανάλογα με το αν βγαίνουν οι δημοκρατικοί ή οι ε, ρεπουμπλικάνοι. Παράδειγμα, Τσεχία, Πολωνία, αντιπυραυλική ασπίδα. Η μία κυβέρνηση λέει Α, η άλλη λέει Β. Εμεί τι λέμε οι Ευρωπαίοι. Ποια είναι η εξωτερική μα πολιτική, Ποιο είναι ο στόχο μα, Δεν είναι να ε, καταργηθεί για να καταστραφεί όλο το οπλοστάσιο τον όπλο μαζική καταστροφής. Για τον αφοπλισμό τι λέμε θα πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να βασίζεται σε μια αυτόνομη, ξεκάθαρη πολιτική που να έχει και ρόλο και χώρο στη διεθνή πολιτική, που να βασίζεται στο βασικό στόχο του αφοπλισμού, του πλήρους όμως αφοπλισμού. Θυμάστε τον Ούλοφ με τον Βίλι Μπραντ κτλ. Όταν ήταν ακόμα οι συνασπισμοί θα πρέπει να έχουμε μια εξωτερική πολιτική που να ακολουθεί αυτό το στόχο και να είναι προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο και να μην στρατιωτικοποιούμε την ασφάλειά μας, που είναι πάγιες συστάσεις της Λισαβόνας, της συνθήκης. Εν πάση περιπτώσει, κυρίε και κύριοι, εμεί ε, παίρνουμε τι αποστάσει μα πλήρω από του ευρωσκεπτικιστέ. Δεν είμαστε σε αυτό το δρόμο. Είμαστε υπέρ τη Ευρώπη, αλλά είμαστε ευρωαπαιτητικοί, επαναλαμβάνω. Και όχι ευρωσκεπτικιστέ. Όλα αυτά που προτείνονται ω αρχιτεκτονική δεν νομίζω ότι είναι η διαδικασία που μα επιτρέπει να φτάσουμε στο παλιό όραμα του Βίκτορο Ουγγό, του 1848 των ε, Ευρωπαϊκών Ομοσπονδών Κρατών. Πάμε σε άλλη κατεύθυνση σε περίπτωση που ε, κυρωθεί, αν κυρωθεί στις χώρες που δεν έχουν κυρώσει ακόμα και παραμονές και αναμένοντας και τη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί φαίνεται και συντηρητική ε, στο συνέδριό τους ε, το έχουν κάνει και αυτό ζήτημα. Επαναλαμβάνω, εμεί είμαστε απαιτητικοί, όχι σκεπτικιστέ και τελειώνω με την κριτική και πάλι προ την γραμματεία. Δεν μπορείτε να μα φαίνετε χτε ένα έγγραφο και να μα λέτε αύριο λίγη, ξέρετε, η προθεσμία για την κατάσταση των απολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση αυτή. Λούνατσεκ. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μέγερ. Εσείς πολύ σωστά είπατε ότι είσαστε της ε, ΓΚΟΕ και είσαστε απαιτητικοί. Δεν είσαστε ευρωσκεπτιστικές. Ε, αλλά και εμείς οι πράσινοι είμαστε πολύ απαιτητικοί. Δηλαδή θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που μας ε, δίνει η συνθήκη. Και τώρα που ψήφισε η Ιρλανδία υπέρ, αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον μπορούμε να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Ξέρω ότι εσείς δεν έχετε την ίδια γνώμη αλλά θεωρώ ότι με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας θα έχουμε περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη και το Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερα δικαιώματα. Γι' αυτό με εκπλήσει κάπως εσείς που είσαστε ευρωβουλευτές δεν τάσεστε υπέρ της συνθήκης, αλλά αυτό το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συζητήσει αλλού. Τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Χάρηκα ιδιαίτερα το Σάββατο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ε, Ιρλανδία γιατί πραγματικά είναι σαφές ότι για δεύτερη φορά οι Ιρλανδοί με μια πλειοψηφία των δύο τρίτων είπαν ναι στην ε, αύξηση, επέκταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Και βεβαίως εγώ θέλησα ε, να στηρίξω τους πράσινους της Ιρλανδίας και πιστεύω η μεγάλη διαφορά με την πρώτη φορά είναι ότι αυτή τη φορά οι θεσμοί, όπως ε, παραδείγματος χάρη τα συνδικάτα, έλαβαν το θέμα πολύ σοβαρά. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά όπου το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ε, υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό δεν εμφανίστηκε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι μερικές ε, φορές Υπάρχει ένα εκνευριστικό, παράλογο επιχείρημα που παρουσιάστηκε από μερικές ομάδες, αυτή τη στιγμή όμως εξαφανίστηκε. Και μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αν δει κανείς τη συνθήκη ε, θα δει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Παραδείγματο χάρη ένα επιχείρημα σχετικά με τον ελάχιστο μισθό που θα κατέβει στο 1,84 με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εγώ σκέφτηκα, μα ποιος μπορεί να λέει όλα αυτά. Όμως, ξέρετε κάτι, ε, ήταν κάτι που υπήρχε σε αφήσει ε, στο Δουβλίνο που έλεγε ότι το ελάχιστο, ο ελάχιστος μισθός θα πάει στο 1,84. Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά ε, δεν τα πίστεψαν και πολλοί άνθρωποι και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής. Όπως σας είπα προηγουμένως, το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν εκείνοι που τάσσονται υπέρ της ε, συνθήκης και το να ανήκει κανείς ε, σε αυτήν την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Υπήρξαν πολλοί νέοι που έκανε εκλογική εκστρατεία υπέρ της συνθήκης. Ε, το βασικό επιχείρημα είναι πού ανήκουμε τελικά, γνωρίζοντας βέβαια ότι και η οικονομική κρίση ε, κάνει στους ανθρώπους να προβληματίζονται. Εγώ θεωρώ ότι ε, υπάρχει αυτό το συνέστημα του που ανήκουμε, ακόμα και αν δεν μας αρέσει. Βεβαίως και πολλοί επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει τώρα και επιθυμούν να βελτιωθεί. Όσον αφορά τώρα το τι θα κάνουμε στο μέλλον, ορισμένοι συναδελφοί μου ήδη μίλησαν Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Κασίνσκι είπε ότι θα ψηφίσει και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Με τον κύριο Κλάους ε, υπάρχει ακόμα κάποιος δρόμος και πιστεύω ότι υπάρχουν εδώ αρκετοί που έχουν καλές επαφές μαζί του και μπορούν ίσως να τον επηρεάσουν, να υπογράψει. Δύσκολο βέβαια. Όσον αφορά τον κύριο Κάμερον ε, και τους συντηρητικούς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εγώ, ε, κοιτάξτε, ήμουνα ε, το Σαββατοκύριακο στην Αγγλία και παρακολούθησα λιγάκι τηλεόραση. Και εγώ λοιπόν έχω την εντύπωση από το συνέδριο των συντηρητικών ότι ο κύριος, ε, το, κύριος Κάμερον τα μαζεύει λιγάκι. Και λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πειράσω κανέναν άλλον αρχηγό κράτους σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση του κυρίου Κάμερον, αυτή είναι κάτι που αν δεν τα μαζέψει δεν θα αρέσει στους συντηρητικούς. Ο κύριος ε, ε, Μπρόκ ε, παρουσίασε μια κατάσταση και αυτό που είπε σχετικά με την αντιπολίτευση πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς θα το πάρουν στην Αγγλία. Τώρα, ε, κατά τα άλλα, πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση πέρα από τον εκδημοκρατισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, είναι σημαντικό να έχει κανείς κατά νου τους πολίτες. Η πρωτοβουλία των πολιτών, κυρίως σε κάποιες χώρες ε, όπου υπάρχει ευρωσκεπτικισμός, όπως είναι η δική μου χώρα, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν ε, τα πράγματα μέσα από τις πρωτοβουλίες τους. Και υπάρχει ένα πράγμα που ελπίζω για την εξωτερική πολιτική και για το ρόλο που θα παίζει η Ευρώπη στον κόσμο, να είναι πιο ισχυρή η Ευρώπη και κυρίως να υπάρχει μια ισχυρότερη φωνή για τα θέματα που υπερασπιζόμεθα και εγώ προσωπικά, ανθρώπινα δικαιώματα, πρόληψη συγκρούσεων και αυτό αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Ε, η πρόληψη ε, των συγκρούσεων είναι κάτι επί το οποίο και το Κοινοβούλιο πρέπει να στρέψει την προσοχή του. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα ε, και θέλω να πιστεύω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε υποστήριξη για όλα τα θέματα έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά να προβληθούν. Al eh, collega Pöttering. Ο κύριος Πέτερνγκ έχει το λόγο. Um Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να ε, πω κάτι σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Νάιτς. Και πριν ε, πω αυτά που έχω κατά νου, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτά που είπε ο ε, κύριος Μπροκ σχετικά με την τον αρχηγό τη αντιπολίτευση στη Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει κανεί να έχει κατά νου την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπο αυτό θέλει να αποσύρει το λόγο που έχει δώσει η Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, συμφώνησαν οι δύο βουλέ, ε, υπέγραψε η Βασίλισσα, η συνθήκη έχει κατατεθεί στη Ρώμη και τώρα θέλει δημοψήφισμα. Αυτό όμω σημαίνει ότι δεν τηρεί το λόγο του και η δέσμευση της Μεγάλης Βρετανίας αποσύρεται. Και αν είναι αλήθεια ότι το άτομο αυτό κάλεσε τον πρόεδρο της Τσεχίας να μην υπογράψει, αυτό κατ' ουσίαν είναι ε, ανατρεπτική ε, στάση. Λέει σε έναν πρόεδρο να μην τηρήσει το Σύνταγμα. Για σκεφτείτε ένας ε, άλλος ε, Ευρωπαίος θα έκανε αυτό που κάνει ο πρόεδρος της Βρετανίας. Ξέρω βέβαια ότι κατά κανόνα εγώ είμαι πολύ προσεκτικός ε, στη διατύπωση που επιλέγω, αλλά το πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος αυτό, αυτός δεν είναι μόνο παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά είναι και μια μορφή υπεριαλισμού, διότι ε, οι 27 χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο και μόνο επειδή καθυστερεί μια υπογραφή, είναι όμοιροι καταστάσεων. Πρόκειται λοιπόν για παραβίαση του συντάγματος και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με όλα μας τα μέσα. Σχετικά τώρα με αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Νάιτς, αγαπητοί συνάδελφε, έχω μία παράκληση. Την ε, τοποθέτησες, την βρίσκω πάρα πολύ καλή, όμως ως Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνουμε στη διπλωματική υπηρεσία να... δεν έχετε μετάφραση. Όχι, καταλαβαίνει γερμανικά. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, εγώ ακόμα δεν είχα τη δυνατότητα να σας μιλήσω για τη διπλωματική υπηρεσία, να παρουσιάσω το δικό μου το κείμενο. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να σας πω. Κοιτάξτε, εγώ από αυτά που είπατε κατάλαβα ότι είχατε τοποθετηθεί. Έκανα λάθος τέλος πάντων. Ε, ίσως μπορώ να πω κάτι και ίσως μπορεί να το λάβει υπόψη συνάδελφος κυρία Νάιτς. Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το κείμενο αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ θέλω να παρακαλέσω στο κείμενο να συμπεριλάβουμε μία διατύπωση έτσι ώστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται σε αυτή τη διπλωματική υπηρεσία. Να μην εξαιρούμεθα, διότι ε, χρειαζόμεθα να συμμετέχουμε σε ε, σημαντικές αντιπροσωπείες και αν δεν το επιτύχουμε εκ των προτέρων, εκ των υστέρων θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν η Στάντος κυρία που θα μιλήσει τώρα εντός λίγο, παρακαλώ να το λάβει υπόψη αυτό που λέω δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται στις ε, διεθνείς εκπροσωπήσεις, στις αντιπροσωπήσεις αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που παρεμβαίνουν να παραμένουν στο πρώτο τμήμα, δηλαδή ως προς την επιτυχία του δημοψηφίσματος, στο γενικό, στην γενική εμβέλεια του θέματος και μετά η συγγήτρια θα μας ε, μιλήσει τις ε, θεσμικές ε, πτυχές σε σχέση με την ευρωπαϊκή εξωτερική δράση, με το ρέλεξ. Θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Κόμματσεφ. Много Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και πολλοί προαρίσαντες, χαίρομαι πάρα πολύ από το αποτέλεσμα ε, της Παρασκευής και του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφεραν οι Ιρλανδοί πολίτες να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στη στάση που έχουν απέναντι στην ίδια τους την κυβέρνηση και στη στάση που έχουν απέναντι στην Ευρώπη που χρειάζεται ένα όραμα και ένα νέο κείμενο μεταρρυθμιστικής συνθήκης και μέσω κρίσης. Βέβαια, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι έπαιξε ρόλο και η κρίση, όντως, ε, ε, το αποτέλεσμα αυτό. Αν δεν ήταν μέρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία θα είχε υποστεί τόσο βαρύ πνίγμα όσο και η Ισλανδία, η οποία τώρα ζητάει να μπει στην Ένωση. Κατά τα άλλα, εγώ όμω δεν συμφωνώ να δίνονται ιδιαίτερα προνόμια σε κάποια κράτη-μέλη για να συμφωνούν με την Α Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Δεν μ' αρέσει αυτό όπως είναι τα προνόμια τα φορολογικά ή τα κοινωνικά που δόθηκαν στην Ιρλανδία. Η συνθήκη της Λισαβόνα σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε ρυθμίσεις ε, όπως ισχυρίστηκαν ε, οι υποστηρικτές του όχι στην ιρλανδια η συνθηκη της λισαβονας σε καμια περιπτωση δεν υποχρεωνει τα κρατη μελη Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αν θα συσταθεί με βάση τη συνθήκη της Νίκης ή της Λισαβόνας. Από ό,τι κατάλαβα, ο πρόεδρος Βαρόσο προτίθεται να περιμένει λίγο για να κάνουν ε, τις προτάσεις και να πάρουν τις αποφάσεις του στα κράτη-μέλη για το πώς θα προχωρήσουν. θα χαιρόμουν πάρα πολύ ε, αν μπορούσαν να μας πούν δύο λόγια οι Πολωνοί, οι Τσέχοι, οι παρόντες συνάδελφοι. Είμαι βέβαιος ότι ο Πολωνός πρόεδρος σε λίγες μέρες θα υπογράψει σε ό,τι αφορά τώρα τις απόπειρες στην τσεχική δημοκρατία να αποτραπεί η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, είμαι βέβαιος ότι θα αποτύχουν οι απόπειρες αυτές και θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη το συντομότερο για να μπορέσει να ε, συσταθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Νέιτς, θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία, η Διπλωματική Υπηρεσία. Θα ξαναπάρω το λόγο μετά για να σας πω τι έχω να σας πω και γι' αυτό. Εμείς έχουμε λάβει μια γνωμοδότηση τώρα. Αυτή η γνωμοδότηση που βασίζεται. Σε πρωτοβουλία της Επιτροπής μας τι είδους γνωμοδότηση είναι αυτή, πώς ορίζεται. Ποια ε, θα είναι η κριτική μας απέναντι στην υπηρεσία αυτή στον Ήπατο. Μα η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι αρμόδια επί της ουσίας. Εμείς γνωμοδοτούμε. Prego, la parola al collega Vigenin, o Vigenin. Vigenin.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 ε, θα μπορούσαμε να ακούσουμε πώς θα ε, προωθηθεί το θέμα της εξωτερικής κοινοτικής ε, δράσης από την υπεύθυνη, από την εισηγήτρια. Εμείς οι σοσιαλιστές και δημοκράτες χαιρόμαστε με την θετική έκβαση την τελική έκβαση. Όπως ξέρετε, είχαμε προωθήσει μία εκστρατεία κατά πρώτη, το πρώτο δημοψήφισμα και τώρα χαιρόμαστε που το δεύτερο στέφθηκε από επιτυχία. Νομίζω ότι η έκβαση θα έχει ε, μεγάλες επιπτώσεις στο, στην εξωτερική και εσωτερική δράση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ναι της Ιρλανδίας θα θέσει τέλος στη θεσμική κρίση και τις ε, αβεβαιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να έχουμε μία πιο δυνατή ε, εικόνα προς, το, προς τα έξω. Βεβαίως έχουμε το θέμα της κύριος από τους Πολωνούς και τους ε, Τσέχους. Χαίρομαι διότι ο Πολωνός Πρόεδρος ε, είπε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει, δηλαδή να κυρωθεί η συνθήκη από την Πολωνία και πιστεύω ε, γνωρίζετε ότι, γνωρίζετε πώς κινείται ο Τσέχος πρόεδρος. Αν τον πιέσουμε υπερβολικά, ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθεί θετικά, αλλά τη στιγμή που ο Πολωνός ε, πρόεδρος κυρώσει τη συνθήκη, τότε θα έχουμε ένα μόνο πρόεδρο που θα αντιτάσσεται στην συνθήκη της Λισαβόνας και εάν οι Τσέχοι δεν κυρώσουν, τότε το θέμα θα σχετίζεται με το συγκεκριμένο άτομο, τον πρόεδρο, αλλά και με ολόκληρη την τσεχική δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην τσεχική δημοκρατία που τάσσονται υπέρ της συνθήκης της ε, Λισαβόνας θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουμε τον Πρόεδρο είναι εσωτερικό θέμα και νομίζω ότι και τα δύο σώματα έχουν κυρώσει και η Γερουσία και η Βουλή, άρα δεν μπορούμε να πιέσουμε περαιτέρω. Γνωρίζουμε το αξιοπερίεργο του χαρακτήρα του Προέδρου της Τσεχίας και αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Επίσης, η Βρετανή συντηρητική θα πρέπει να είναι σαφής. Αυτές οι φήμες ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Τσέχου Προέδρου και του Ντέιβιτ Κάμερον ότι οι Τσέχοι θα απαγώσουν την ε, συνθήκη, την κύρωση δηλαδή έως ότου κερδίσουν εκλογές οι συντηρητικοί, μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα ε, δεν υπάρχει μία ε, σοβαρή πολιτική ε, ανταπόκριση και βάση περιπτώσει δεν είμαστε και σίγουροι ότι οι του χρόνου θα κυβερνήσουν στη Μεγάλη Βρετανία. Και δεν νομίζω ότι θα είχαν τόσο περίεργη πολιτική συμπεριφορά. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα γίνει η κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Υπάρχουν και ορισμένα επιπρόσθετα θεσμικά ζητήματα και θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε μάλλον μέχρι ότου έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η άποψη της σοσιαλιστικής ομάδας είναι ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε μία νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναμη της συνθήκης της Λισαβόνας όταν κυρωθεί από όλους. Βεβαίως θα συνεχίσουμε με την προπαρασκευή της ψηφοφορίας για την επόμενη Επιτροπή τους ε, κανόνες που ισχύουν τώρα, αλλά θα θέλαμε να γίνει η εκλογή δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Βεβαίως υπάρχει και ένα ε, ερωτηματικό προς την εκλογή του Πρόεδρου Μπαρόζο, διότι η εκλογή έγινε δυνάμει της συνθήκης της Νίκαιας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε έναν πρόεδρο που εξελέγει δυνάμει της συνθήκης της Νίκαιας και ολόκληρο το διευθυντήριο τους επιτρόπους δηλαδή που εκλέγονται δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας μην το θεωρήσετε προκλητικό αλλά ίσως θα μπορούσε να γίνει και μια νέα ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης νομική διαφάνεια επί του θέματος. Τέλος, νομίζω ότι τη στιγμή που θα κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας το Συμβούλιο και ο ίδιος ο Μπαρόζο θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να είναι ή μάλλον θα είναι υπεύθυνη, ιδιαίτερα υπεύθυνη για το, τον πρώτο πρόεδρο του Συμβουλίου και τον είπα το εκπρόσωπο, ως προς το ρόλο αυτών των δύο προσώπων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τη στιγμή που υπάρχει νομική βάση για τα δύο αυτά πρόσωπα και τη στιγμή που θα ξέρουμε ποια θα είναι και τα πρόσωπα αυτά, Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική θα πρέπει να εκπροσωπεί το σοσιαλιστικό κίνημα έτσι ώστε να γίνει σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στην όλη διαδικασία για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ως προς τις ε, θεσμικές πτυχές. Ε, με βάση την ε, θέση της εισηγήτριας και αυτή θα είναι και η αρχή. Διότι υπάρχουν πολλές ε, προκλήσεις σε σχέση με την ΚΕΠΑ για το μέλλον και τώρα θα πρέπει να επηρεάσουμε τη διαδικασία εφόσον πρόκειται για μία νέα αρχή θα πρέπει να διαμορφώσουμε την κατάσταση υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών έτσι ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν τον σημαντικό ρόλο που τους αρμόζει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κασουλίδης, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο λαός της Ιρλανδίας είναι κυρίαρχος λαός, ψήφισε ναι και ήταν κυρίαρχο, κυριαρχικό το δικαίωμα να ψηφίσει διαφορετικά από την περασμένη φορά. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά ψήφισαν ναι, διότι το Συμβούλιο δεσμεύτηκε ρητά για ζητήματα που την τελευταία φορά τους οδήγησαν να ψηφίσουν όχι. Παρά το γεγονός ότι όλα τα ζητήματα της δέσμευσης δεν ήταν θέματα που αφορούσαν τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά η εκστρατεία του όχι προσπάθησε να παραπλανήσει το λαό προς την κατεύθυνση αυτή. Και ας μην λησμονούμε και πάλι ότι στο μεταξύ ε, μεσολάβησε και η οικονομική κρίση και η χρηματοπιστωτική που έδειξε πόσο αλληλεπίδραση, πόση αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ όλων μας και πόσο κρίσιμο είναι να ανήκει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνούμε και την περίπτωση της Ισλανδίας που δεν ήθελε να μπει στην Ένωση και τώρα είναι υποψήφια χώρα ακριβώς λόγω όλων ε, αυτών που υπέφερε ως μικρή χώρα από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Μικρή χώρα με μικρό νόμισμα που δεν μπορούσε να αντέξει τις διεθνείς πιέσεις. Άκουσα το επιχείρημα ότι ο λαός της Ιρλανδίας λέει θα έπρεπε να ψηφίζει ξανά και ξανά μέχρι να πέρασει το ναι. Γιατί στο Ηνωμένο όχι συγγνώμη, το πω ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι προσπαθούν να κάνουν οι συντηρητικοί. Ακριβώ το ίδιο. Ε, και αυτό το λέω προ εκείνου που χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα. Ε, στη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και με την υπογραφή της Βασιλίσης έχει επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνα και τώρα κάποιος προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να αλλάξει γνώμη. Μα είναι προφανές ότι πολλοί από εμά υποτιμούμε ε, τη εστί αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εμείς συζητούμε εδώ ε, στο Κοινοβούλιο ως εκπρόσωποι ακριβώς αυτής της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν με αυτόν τον τρόπο κυρώσει τη συνθήκη που ε, είναι εξίσου έγκυρη μέθοδος όσο το δημοψήφισμα. Και ξέρουμε ότι σε περίπτωση δημοψηφίσματος ε, μπαίνουν πολλά ζητήματα άσχετα τελείως με το αντικείμενο του δημοψηφίσματος. Και γι' αυτό μερικές φορές έχουμε αποτελέσματα που δεν έχουν καμία σχέση με το ερώτημα που ετέθη. I want to say that I was Πρέπει να σας πω ότι ένιωσα ανακούφιση από κάποιες δηλώσεις του Προέδρου Βάκλαφ Κλάους στη Πράγα γιατί νομίζω ότι έστειλε το μήνυμα προς τους Βρετανούς συντηρητικούς ότι είναι πολύ αργά πλέον για να περιμένουν ότι μπορεί αυτός να καθυστερήσει μέχρι το, να γίνουν εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μην υπογράφει. Ε, ε, είναι λογικό αυτό και είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος είναι πολύ εχέφρον άνθρωπος και γνωρίζει ότι ε, ποιο είναι το επιχείρημα και η θέση του συνταγματικού δικαστηρίου. Έχουν προσφύγει πολλοί σε δικαστήρια συνταγματικά και στο γερμανικό και στο τσεχικό ε, και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να υπάρξει νέα απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου και να μπορέσει να υπογράψει να υποχρεωθεί να υπογράψει τη συνθήκη της Λισαβόνα. για να τεθεί πλέον σε ισχύ μέχρι την αρχή του επομένου έτους. Αυτή στιγμή τώρα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνα. και γίνει νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελειώνω με αυτό πρόεδρε, τότε δεν θα μπορεί μία και μόνη χώρα να ε, κρατάει όμοιρο της απόφασης της. Το αντίστροφο θα γίνει. Λοιπόν, οι τόριδες να τα ακούν αυτά γιατί αν ε, σκοπεύουν να κάνουν διάφορα, ε, εκείνοι θα πρέπει να πείσουν τους 27, 26 υπολείπους. Και σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Βίγκενιν για τον κύριο Μπαρόσο, αυτό το ζήτημα νομίζω έχει λυθεί. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελήφθη διαπαντός αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα νομιμότητας. διότι έλαβε και την πλειοψηφία που απαιτεί συνθήκη της Λισαβόνας, ξέρετε. Και αν η ε, νομιμότητα ε, τη εκλογής του κυρίου Μπαρόσο τεθεί ένα του, θα πρέπει κανείς να αμφιβάλλει και για την ομότητα του Κοινοβουλίου μας, που επίσης εξελέγει με βάση τη συνθήκη της νίκαια. Έχουμε τρεις τελευταίες παρεμβάσει. Θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα ε, συνεκτικοί πριν λάβει το λόγο ο εισηγητή. Λούλινγκ. Α, Λουέζινγκ, με συγχωρείτε. Ja, Dank. Ευχαριστώ, κυρία Λόζενκ. Πολλά ακούστηκαν σήμερα για τη δημοκρατία στη Γερμανία. Ε, λένε οι άνθρωποι ε, της ε, αγοράς και του εμπορίου όταν κάτι δεν μας ταιριάζει, το, ταιριάζουμε εμείς. Ε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ για τη δημοκρατία. Η ελευθερία της γνώμης, τα δημοψηφίσματα, η συναπόφαση, όλα αυτά είναι δημοκρατικές έννοιες πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά η δημοκρατία είναι δύσκολο οικοδόμημα. Ε, στην Ιταλία είχαμε ε, διαδηλώσεις για την έκφραση γνώμης. Προφανώς δεν θα ε, απαγορεύεται δια νόμου ε, στην Ιταλία, αλλά το θέμα της ελευθερίας της γνώμης έχει να κάνει με ποιο κατέχει τα μέσα και τη γνώμη. Και πραγματικά έχουμε ε, παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων. Ερωτώ, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άραγε υποχρεωμένα σε τέτοιες διαδικασίες ε, όπως είναι τα δημοψηφίσματα των λαών να τηρούν στάση ουδετερότητας. Το αντίθετο, πήγανε πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία για να συμμετέχουν στην εκστρατεία υπέρ του ναι. Χρησιμοποίησαν κονδύλια που παραβιάζουν ε, το Ιρλανδικό δίκαιο και κυβερνητικά κονδύλια και άλλα κονδύλια που χρησιμοποίησαν και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ναι. Εταιρείε το έκαναν. Εντάξει, επιτρέπεται, αλλά είναι δημοκρατικό και αυτό. Που ε, ε, επένδυσαν ε, χιλιάδες σε αυτή την εκστρατεία του ναι. Και επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Είναι άραγε όλα αυτά δημοκρατικά και είναι και νόμιμα. να πηγαίνουν εκπρόσωποι και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζικά ε, και να συμμετέχουν ε, στη δημιουργία γνώμης ε, και στη διαμόρφωση της γνώμης ενός ολόκληρου λαού. Ο συνάδελφος Μπροκ είπε ότι υπήρξε και μεγάλη κατασυκοφάντηση και υπάρχει κατά της συνθήκης. Γενικά επενούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα έχει μεγαλύτερη συναπόφαση. Ερωτώ, ε, ουσιαστική συναπόφαση θα έχει για να στέλνουμε στρατιώτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στο άρθρο 36 δεν βρήκα ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το δικαστήριο στο 275 έχουν δικαίωμα λόγου ουσιαστικό. Σε περίπτωση πολέμου και ειρήνης η διάκριση των εξουσιών κατ' εμέ ε, έχει καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα με ενδιαφέρει πολύ και η δική σας γνώμη. Αυτά και σταματώ. Και μετά ο κύριος ε, Πρέντα. Για το... Και μετά θα εκφραστεί η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα... Να... Ε, ήθελα να σας πω ότι συμμετείχα στην ε, σύνταξη στη σύνταξη του, της κύρωσης, του κειμένου κύρωσης ε, και θα ήθελα να σας πω, συνάδελφοι, σήμερα ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας θα κυρώσει τη συνθήκη στο εγγύς μέλλον, το πιστεύω αυτό και νομίζω ότι θα επισυμβεί πολύ σύντομα. Τότε στην Πολωνία ε, θεώρησα ότι η διαδικασία δεν θα είναι καθόλου εύκολη, όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, όπου ανέκυψαν πολλά επιμέρους ζητήματα. Νομίζω ότι τα καλά νέα από το Ιρλανδικό δημοψήφισμα είναι ότι τώρα έχουμε μία ουσιαστική δημόσια συζήτηση στα κρατη Μία δημόσια συζήτηση ως προς το θέμα της συνθήκης και το περιεχόμενο της συνθήκης. Η συνθήκη δεν είναι τόσο καλή όσο την θέτουν οι υπέρμαχοί της, αλλά δεν είναι και τόσο κακή όσο ε, ορίζουν οι αντιφρονούντες, ας το πούμε. Υπάρχει διαδικασία συνεργασίας που προβλέπεται σε πολύ δυσχερείς καταστάσεις ε, υπό τη θεσμική έννοια η συνθήκη αποτελεί και επιτελεί πρόοδο, διότι προβλέπει θεσμικά όργανα που θα βοηθήσουν την Ένωση να λειτουργήσει πιο σωστά, δηλαδή τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Αλλά ποιος θα είναι ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου. Θα είναι ένας ρυθμιστής ή θα είναι ένας νέος ατύλας ένας ατήλας, όχι νέος, ένας ατήλας. Και υπό το φως ε, αυτής της επιλογής, ποιος θα είναι και ο ρόλος του Συμβουλίου, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου όπως προβλέπετε. Επίσης, η συνθήκη ορίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εξωτερικές σχέσεις πολλά, μάλλον μερικά συνταγματικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί επί της συνθήκης σε ορισμένα κράτη-μέλη και θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στην πρώτη απόφαση της τσεχικής δημοκρατίας αλλά και την ουσιαστική απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου της Κάρλς που αναφέρεται στο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και το συσχετισμό, τη διάδραση που θα υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια της ε, επικουρικότητας γίνεται όλο ένα και πιο σημαντική και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτό το σώμα θα ορίσει αυτές τις καλώς διαρθρωμένες σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όπως ξέρετε, ε, ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων στο Εθνικό μου Κοινοβούλιο και γι' αυτό με ενδιέφεραν οι θεσμικοί αυτοί οι συσχετισμοί, γιατί δεν θα επιθυμούσαμε τα εθνικά κοινοβούλια να θεωρήσουν ότι η γνώμη τους δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Άρα δεν εκμεταλλευόμαστε τις συνθήκες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ως προς την, ε, τη λειτουργία της Ένωσης, δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας, Εδώ μπορώ να πω ότι όλα θα εξαρτηθούν θεσμικά από τη ε, δυνατότητα συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων δεν μπορεί αυτό να το ορίσει επακριβώς μια συνθήκη. Όλα εξαρτώνται από την καλή θέληση όλων. Και η βρετανική εμπειρία είναι σωτήρια. Διότι είδαμε την κύρωση η οποία ε, ίσχυσε, αλλά τώρα αμφισβητείται. Ο συνάδελφος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω την χαρά μου για την καλή έκφαση του ε, δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας. Θα ήθελα όμως να παρατηρήσω ότι είναι γεγονός ότι η επανάληψη ενός δημοψηφίσματος δεν δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης, διότι δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε πάντα ότι οδηγεί στην πραγματική εμπιστοσύνη των πολιτών. Νομίζω ότι οι λόγοι αυτής της εμπιστοσύνης σχετίζονται με διαφανή αποτελέσματα. Εάν το αποτέλεσμα ε, ήταν ε, γύρω στο 50% τότε θα υπήρχε μεγαλύτερη αναποφασιστικότητα. Το 67% όμως αύξησε την εμπιστοσύνη. Ο κύριος Γκρίς μίλησε για την κατάσταση στην Πολωνία και ελπίζω η Πολωνία να μην αργήσει να κυρώσει όπως υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Πολωνίας και θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λούνατσεκ ότι δηλαδή τα κόμματα έχουν λάβει πολύ στα σοβαρά το θέμα, το θέμα της συνθήκης. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά έχει καταβληθεί αυτή η προσπάθεια και έχει επιβληθεί αυτό το αποτέλεσμα εξαιτίας της ε, κρίσης. Δηλαδή, αυτά τα πολιτικά αποτελέσματα είναι απότοκα μιας κατάστασης ε, κρίσης και είναι πολύ δύσκολο πάντα να προχωρήσει η Ευρώπη σε συνθήκες ε, κρίσης. Όμως ο πρόεδρος της ε, Τσεχίας συντάχθηκε με δυνάμεις της αντιπολίτευσης, διότι ο κύριος ε, Κάμερον δεν βρίσκεται στην ε, κυβέρνηση. Μάλλον το κόμμα του δεν είναι κυβερνών κόμμα και θα ήταν περίεργο, αξιοπερίεργο να έχει συμφωνήσει με έναν ενδεχόμενα μελλοντικό πρωθυπουργό ο Τσέχος πρόεδρος, δηλαδή με τον κύριο ε, Κάμερον. Ως προς αυτά που είπε ο κύριος ε, ε, Βινέγκιν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα ιδιαίτερα στρεβλωτικό αποτέλεσμα και ελπίζω να μην ισχύσει αυτό για την Μεγάλη Βρετανία. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Βιγγένιν όμως ως προς την εκλογή του Πρόεδρου Μπαρόζου, γιατί πιστεύω ότι ήταν απόλυτα νόμιμη η εκλογή του κύριε Βιγγένιν και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τεθεί ένα αμφιβόλο. Αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για το σχέδιο γνωμοδότησης η κυρία Νέιτς έχει το λόγο, η συγγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Επιτέλους λοιπόν μου προσφέρεται η ευκαιρία να παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να σας πω ότι έγιναν κάποιες ε, παρατηρήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζω βέβαια ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ πολύ περιοριστικό και οφείλεται στο εξή. Ο συνάδελφος κύριος Μπροκ ε, εργάστηκε για το σχέδιο της ε, εκθεσής του και νομίζω επίσης ότι η συνδιάσκεψη των Προέδρων αυτού του Κοινοβουλίου αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Να αναβάλει τη συζήτηση μέχρι να γνωρίζουμε ακριβώς ε, το αποτέλεσμα του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Το Ιρλανδικό λοιπόν δημοψήφισμα έλαβε χώρα την Παρασκευή και ως εκ τούτου Συζητήσαμε την έκθεση του κυρίου Μπρόκ σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και τώρα συζητάμε τη δική μου τη γνωμοδότηση σε αυτήν την Επιτροπή. Όμως ε, αποφασίσαμε από κοινού με τη γραμματεία που παρεπιπτόντως δεν ευθύνονται για αυτές τις ε, ημερομηνίες, γιατί αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουμε. Ως εκ τούτου είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί ευθύνονται για το ότι το κείμενο διανεμήθηκε με τέτοια καθυστέρηση. Απλά αποφασίσαμε να μην καταθέσουμε κείμενο μέχρι να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, στην Ιρλανδία. Με πάση περιπτώσει, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών μετακινήθηκε, δεν είναι αύριο, είναι στις 8 Οκτωβρίου 5η μεσημέρι. Έτσι λοιπόν έχουμε λίγο χρόνο περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά. Αυτά σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Και στις δύο επιτροπές ε, είμαστε ε, δεσμευμένοι να αποφασίσουμε τη Δευτέρα στην Επιτροπή και λίγες μέρες αργότερα πάλι στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια γιατί θέλουμε να λάβουν χώρα αυτές οι ψηφορίες ε, την επόμενη φορά στο Στρασβούργο, διότι τα κείμενα θα είναι έτοιμα και ε, θα κατατεθούν πριν από την άτυπη συνάντηση που θα λάβει χώρα λίγες μέρες αργότερα. Όπως γνωρίζετε, η Σουηδική Προεδρία επιθυμεί να συνεχίσει με όλες τις συζητήσεις για το θέμα αυτό για την ε, ε, κατανομή θέσεων ε, τον Ευρωπαίο Πρόεδρο, τον είπα το εκπρόσωπο και το καθεξής. Όλοι λοιπόν θεωρούν ότι οι συζητήσεις αυτές θα αρχίσουν σοβαρά στην άτυπη συνάντηση κορυφή. Εμεί επιθυμούμε η δική μα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι έτοιμη πριν ξεκινήσουν. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει τέτοια πίεση χρόνου. Γνωρίζω βέβαια ότι δεν βολεύουν όλα αυτά. Ελπίζω όμω να κατανοείτε τα πολιτικά αίτια που μας οδήγησαν στο να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά τη γνωμοδότησή μου, ξεκινάει με κάποιες γενικές παρατηρήσει, όπου βέβαια ε, καλωσορίζουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας. Είχαμε βάλει στίχημα ότι θα είναι θετικό και γι' αυτό λέμε εδώ χαιρετίζουμε το δημοψήφισμα και το καθεξής. Όσον αφορά τώρα τις αλλαγές ε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, εδώ θέλω να πω μία αλλαγή θα είναι ότι ο ύπατος εκπρόσωπος που θα είναι και αντιπρόεδρος της Κομισιόν θα συνεπικουρείται από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Δράσης, Εξωτερικής Δράσης. Ε, χαιρετίζουμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά τα θέματα που ζήτησε και ζητούσε ανέκαθεν την σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας. Λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ερωτηθεί για τη σύσταση της EAS και όσον αφορά τις συνέπειες από τον προπολογισμό, πιστεύουμε ότι ένας έγκαιρος και ουσιαστικός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καθοριστική σημασίας για να ξεκινήσει αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και για να διασφαλιστεί ότι θα την χάνει και των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Πάμε τώρα στον ύπατο εκπρόσωπο, ο οποίο ε, καλείται να καταθέσει τις ε, προτάσεις του ή τη το συντομότερο δυνατόν. Και επιμένουμε ε, να υπάρχει σεβασμός των εξή αρχών. Πρώτον, θεωρούμε ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να συσταθεί μέσα στο διοικητικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Κομισιόν και να βοηθάει τον υπατορμοστή στην, ΚΕΠΑ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ίσως είναι μια λίγο περίεργη θέση, αλλά κατά την άποψή μου είναι λογική συνέχεια του τρόπου με τον οποίο εκφράζεται η ε, δυτή διαδιακή αυτή λειτουργία που έχει αναλάβει ο ύπατος εκπρόσωπος. Και είναι ακριβώ αυτό που λέει και ο κύριο Έλμαρ Μπρόκ στο σχέδιο της έκθεσής του. Επίσης επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι η υπηρεσία δράσης ε, πρέπει να ασχολείται και με την ε, κοινή εξωτερική πολιτική, με την ΚΕΠΑ και με, ε, με την ΕΠΑ και επιπλέον ο ύπατος αρμοστής θα πρέπει να καταθέσει μία πρόταση για το πώς άλλες πολιτικές θα ε, οργανωθούν ε, σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε υπογραμμίσει την διεύρυνση, το εμπόριο, την ανθρωπιστική βοήθεια αυτά θα αποτελούν ε, σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπογραμμίζουμε επίσης ότι κατά την άποψή μας υπάρχουν πολλοί λόγοι το γιατί θα πρέπει να περιλαμβάνεται η πολιτική ανάπτυξη σε αυτή τη νέα υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουμε ότι οι άλλες ε, πολιτικές ε, όπως το εμπόριο θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να ενταχθούν ε, σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εξάλλου υπογραμμίζουμε ότι η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μονάδες διαχείρισης στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων, ακόμα και το ότι για στρατιωτικές επεμβάσεις η διοίκηση θα πρέπει να είναι διαφορετική από ό,τι στην περίπτωση των πολιτικών υποθέσεων. Επισημαίνουμε ότι οι αναλύσεις που θα γίνονται θα είναι καθοριστικής σημασίας έτσι ώστε να συνεπικουρείται ο ύπατος εκπρόσωπος στο να εκπληρώνει το καθήκον του με έναν τρόπο συνεπή συνεκτικό και να είναι και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε τον είπα το εκπρόσωπο να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα πρόσληψης και επάντρωσης της υπηρεσίας, γιατί η υπηρεσία θα περιλαμβάνει ε, προσωπικό από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να είναι επαγγελματική, θα πρέπει να είναι ε, ικανοποιητικά πρικοδοτημένη και να δείχνει σεβασμό για τις σωστές διαδικασίες επιλογής ε, και με βάση την γεωγραφική ισορροπία. Οι διπλωμάτες των κρατών μελών και το προσωπικό που προέρχονται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν ε, ε, ισόρροπους ρόλους και θα πρέπει να, είναι, να διέπεται το καθεστώς της πόλης από τι ε, ίδιε συνθήκε όπω και των προσωρινών υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σω αυτή η παρατήρηση σα μοιάζει λίγο κοινότοπη, αλλά είναι απαραίτητη. Γιατί για την εύρυθμη λειτουργία μια υπηρεσία, οποιαδήποτε και είναι αυτή, είναι καθοριστική σημασία οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτήν να εργάζονται με βάση του ίδιου όρου και ε, με τον ίδιο μισθό. Οποτεδήποτε αυτό δεν συμβαίνει, δημιουργούνται τριβέ ανταγωνισμό ε, και δημιουργείται κακό κο αρνητικό πνεύμα. Πρέπει λοιπόν να το αποφύγουμε θυσία, γι' αυτό και ε, κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Επόμενο θέμα. Η δημιουργία ενός ε, ικανοποιητικού πνεύματος ε, για να γίνεται και σωστή η εκπαίδευση. Αυτό είναι καθοριστικός στόχος για να επιτευχθεί ο, ο τελικός στόχος που είναι το πλαίσιο μιας διπλωματίες ενοποιημένης όπου θα εκφράζεται εκφράζονται και οι εθνικές ε, διπλωματίες και οι ευρωπαϊκοί. Ο πολιτισμός, τα κοινά προγράμματα κατάρτισης ε, και ένα κοινό ε, διπλωματικό διοντολογικό πλαίσιο είναι απαραίτητα. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία. Στο επόμενο θέμα μιλάμε για το μέλλον των ε, αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα, τις αντιμετωπίζουμε ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ως εκ τούτου οι αντιπροσωπείς αυτές θα πρέπει να υπάγονται στην, στον ύπατο εκπρόσωπο διοικητικά θα πρέπει να ανήκουν στην Επιτροπή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εδώ κατ' ουσίαν προτείνουμε οι, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να μετατραπούν σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να παραμείνουν διοικητικά τουλάχιστον μέσα στο, στις αρμοδιότητες της ε, Κομισιόν να ε, λαμβάνουν ε, βέβαια τις εντολές από τον ύπατο εκπρόσωπο και να υπάγονται σε αυτόν. Ζητάμε ο ύπατος εκπρόσωπος να δεσμευθεί ότι θα ενημερώνει την Επιτροπή μας Ορισμένοι ίσως επιθυμούν εδώ να δουν γενικότερα το Κοινοβούλιο. Πάντως τη δική μας την Επιτροπή για τους ε, διορισμούς ε, που θα κάνει σε υψηλά κλιμάκια και να συμφωνήσει στο ότι ε, θα γίνονται συνεντεύξεις με τους υποψήφιους εφόσον το επιθυμεί η δική μας Επιτροπή. Επίσης ζητάμε από τον ύπατο εκπρόσωπο να δεσμευθεί έτσι ώστε να αναδιαπραγματευτεί την τρέχουσα θεσμική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση σε ευαίσθητα θέματα και άλλα που είναι καθοριστική σημασία για να υπάρχει ε, αγαστή θεσμική συνεργασία. Σημειώνουμε ότι οι αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες θα συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες των κρατών μελών και θα υπάρχει η δυνατότητα μακροπρόθεσμα να προκύψουν ωφέλη καθότι οι αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αναλάβουν και τα προξενία και να ασχολούνται και με θέματα θεωρήσεων και Σέγγεν. Και τέλος, αυτό είναι ένα σημείο όπου η ε, γνωμοδότηση αυτή αποστασιοποιείται από το σχέδιο έκθεση του συνδέλφου κυρίου Μπροκ, ως εκ τούτου σας επισημαίνω ιδιαίτερα αυτό που θέλω να πω τώρα. Τέλος λοιπόν καλούμε την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και τον επόμενο ύπατο εκπρόσωπο να δεσμευθούν ε, για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα αφορά στην σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό να είναι μια δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν οι ασυνέπειες, η διασπάθηση των πόρων ε, και η θεσμική εναρχία. Και τέλος επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να ασκήσουμε τα δημοσιονομικά μας δικαιώματα σε απόλυτη σχέση με αυτούς τους, ε, τις θεσμικές ε, καινοτομίες. Τελικά θέλουμε να πούμε, να επισημάνουμε ότι όλα αυτά παραμένουν υπό τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Αρχής, όπως ακριβώς προβλέπει η συνθήκη. Γιατί αναφέρα αυτό που σας είπα, διότι έχω μια μεγάλη ανησυχία που κατά την άποψή μου ε, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά. Δεν αντιμετωπίστηκε οποτεδήποτε συζητήσαμε για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας. Ότι δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους που δεν εργάζονται απαραίτητα με διπλωματικό καθεστώς, αλλά εργάζονται στις διάφορες γενικές διευθύνσεις, ε, στους ε, φορείς, οι οποίοι με τον ΑΒ τα τρόπο ε, έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, εμείς ε, ζητάμε σταδιακά να ε, επεκταθεί η εξωτερική αυτή υπηρεσία και βεβαίως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να έρθει σε ανταγωνισμό με τις ε, αντιπροσωπείες της ε, Επιτροπής οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Ε, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που διαφωνούν επ' αυτού. Ε, μερικοί τάσσονται υπέρ της προσέγγισης της μεγάλης έκρησης ε, του Big Bang. Όλοι ε, να μπουν σε αυτό που υπάρχει, στις αντιπροσωπείς επιτροπής. Άλλοι λένε πιο ήπια, πιο σταδιακά. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα με τη Γενέβη, με την Νέα Υόρκη, έτσι για να σε αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Και φοβούμε ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξει ανταγωνισμός, θα υπάρξει διασπάθηση πόρων, επικάλυψη εργασιών και δεν είμαι σίγουρη ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Ακόμα και αν βέβαια αναγνωρίζω ότι προφανώς και θα υπάρξει ένα είδος μεγάλης έκρηξης. Θέλω όμως ε, να επισημάνω τον κίνδυνο του να ε, προκύψουν αναταραχές, ανταγωνισμός και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα επίσης και να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής που ε, με συνέδρα με τα μάλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Νέιτς, αγαπητοί συνάδελφοι. Τόνισε η κυρία Νέιτς, και εγώ δεν, θα κάνω παρά κάποια συμπληρωματικά, ε, ότι σεβόμαστε τους Ιρλανδούς πολίτες, αλλά Υπάρχουν και κάποια υψηλά κέντρα στη δίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου που λογαριάζουν διαφορετικά. Η εξωτερική υπηρεσία θα είναι πολύ σημαντική. Είναι ευρύτατη υπηρεσία, ε, εντάσσεται στον Ήπατο, εκπρόσωπο ο οποίος είπαμε ότι είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει να θυμίζουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει το λόγο του. Επιβάλαμε στη ε, συντακτική συνέλευση ότι αποφασίζεται από το Συμβούλιο αυτή η υπηρεσία μετά από πρόταση του ΥΠΑ του εκπροσώπου ε, με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μιλώ για τον εκπρόσωπο τον επόμενο, όχι τον ΙΝ, αυτόν που θα εκλεγεί και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει έκθεση. Αυτά που κάνει η κυρία Νέιτς, ας πούμε, αυτόν τον καιρό είναι η δυνατότητα διαπραγμάτευσης που έχουμε εμείς για τις διαπραγματεύσεις και συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα χρειαστούν συμβιβασμοί για να συμφωνήσουν τα τρία θεσμικά όργανα μοιραία. Αλλά συμφωνώ και με την κυρία Νέιτς που λέει ότι αυτή η εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και διοικητικά και ε, οικονομικά προς τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λένε αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Και ε, η συνθήκη τι λέει, ότι έχει χαρακτήρα ε, sui generis. δεν σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητη. Αλλιώ θα το έγραφε. Ούτε η υπηρεσία είναι agency. Ε, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την υπηρεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και θεσμικά και οικονομικά. Αλλά αυτό το τμήμα λοιπόν ότι θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι έτσι sui generis γιατί έχει διαφορετικές αρμοδιότητες στα ε, πρέσια της εξωτερικής πολιτικής. Ας πούμε για την άμυνα είναι αρμόδιο το Συμβούλιο. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε η υπηρεσία αυτή να είναι υπό την αιγίδα ε, του υπάτου και αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει πιστά να ε, υπηρετεί και το Συμβούλιο και όχι ε, να εντάσσεται στην απλή λειτουργία την κανονική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ας πούμε υπάρχουν θέματα προσωπικού. Εθνικοί εμπειρογνώμονες, τα είπε η κυρία Νέιτς, θα πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι ισχύει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θα έχουμε από το Συμβούλιο, από τα κρατημέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπαλλήλου τριπλής προελεύσεως. Αυτά τα ζητήματα και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ε, μιας νοοτροπίας, ενός σώματος, του ανήκει σε ένα σώμα, esprit de το λένε αυτό στα γαλλικά, ε, θα πρέπει να το δούμε και πώς θα ε, το προάγουμε σε συνεργασία. Καταρχήν συμφωνώ. Και πολλά από όσα προτείνει η κυρία Νέιτς είναι ενίσχυση και ευπρόσδεκτη των όσων έχουμε αποφασίσει και νομίζω θα ε, καταλήξουμε σε μια κοινή θέση με μεγάλη πλειοψηφία. Για να ε, το αποφασίσουμε αυτό το συντομότερο, να μην αφήσουμε το πεδίο ανοιχτό στα άλλα θεσμικά όργανα και ε, ευχαριστώ την Επιτροπή μας και την παρακαλώ να προχωρήσουμε γρήγορα. Γιατί αυτό ε, εκπροσωπεί συμφέροντα του Κοινοβουλίου και κυρίως συμφέροντα της Επιτροπής μας εδώ. Γιατί είναι θέμα κλειδί αν θα λαμβανόμαστε ε, όπως αρμόζει υπόψη στις δυνατότητες ελέγχου που υπάρχουν. Από την ακρόαση με τον ύπατο εκπρόσωπο και το μόνιμο ελέγχο της εξωτερικής υπηρεσίες. Και δεν επιτρέπεται να αφήσουμε κάποια ζητήματα που είναι κοινοτική αρμοδιότητα, ας πούμε, τα προγράμματα των εξωτερικών σχέσεων, ε, να γίνουν de facto διακυβερνητικά. Υπάρχει ιστοδυνικές κοινοβουλευτικός έλεγχος. Δεν μπορούμε ε, να περάσουμε σε θέματα ενιαίας αγοράς, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, γιατί αλλού ασκείται η πολιτική. Τώρα δυστυχώ έφυγε η συμπατριώτησά μου εξ αριστερών που έχει φύγει. Γιατί φαίνεται έχει να πάει και έκανε εργαστήριο τώρα να κάνει και τίποτα, καμία πρακτική δουλειά και, και νόημα. Ich möchte feststellen. Θα ήθελα να διαπιστώσω. Και αυτό είναι απόφαση του, Ευρωπαϊ... του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για να μην υπάρχουν σφάλματα για το ποια στρατιωτική αποστολή θα εγκριθεί, αυτό είναι θέμα του κάθε κράτους μέλους. Και στη χώρα μου υπάρχει επιφύλαξη της βολής, Bundestag. Και, σε περίπτωση, και στο βαθμό που δεν έχει αλλάξει το δίκαιο, θέλω να διαψηφίσω, ε, να, να διαψεύσω συγγνώμη, ε, κατηγορηματικά αυτή την εντύπωση που προσπαθεί να δημιουργήσει το κόμμα της αριστερά στη Γερμανία, τη Λίνκε, ότι ε, στέλνουμε διάφορα στρατεύματα ε, ερήμην του Κοινοβουλίου. Όχι. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέχεται σε ζητήματα οικονομικά και άλλα. Δεν υπάρχουν εδώ χώροι ε, ε, ε, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι μια συντρέχουσα, όπως λέγεται, αρμοδιότητα και δεν θα πρέπει ε, κανένας να μας ε, κατηγορεί, γιατί είναι πραγματικά συκοφαντία και συκοφαντία που ακούστηκε και στην Ιρλανδία και χρειάστηκε να το εξηγήσουμε. Δεν επιτρέπεται να αποχαυνώνεται έτσι ο πολίτης. Ε, και οι αριστεροί συχνά συναισθηματικά μιλάνε για αυτά τα θέματα, αλλά εκπροσωπούν πολιτικές παραδόσεις που δεν εντάσσω στον πυρήνα εγώ της δημοκρατίας. Όποιος έχει ως κόμμα και ιδιαίτερα η Γερμανία αριστερή, όποια έχει τέτοια παράδοση και τέτοια ιστορία δεν δικαιούται δια να ομιλεί και δια να δίνει μαθήματα για δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Νέιτς και κύριε Μπρόκ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή αυτή σα τη σαφήνεια. Τώρα ξέρω πού βρισκόμαστε, ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προχωρήσουμε με αυτή τη γνωμοδότηση θα γίνουν ε, συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο για το μέλλον της ε, διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα, με βάση αυτή την χτεσινή γνωμοδότηση, να τονίσω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς ως προς την εμβέλεια, την ε, νομική οντότητα και τη νομική βάση για να ξέρουμε πώς θα επανδρωθεί. Η κυρία ναι, Νέιτς είπε ότι ορισμένες υπηρεσίες της ΡΕΛΕΞ, όπως η αναπτυξιακή πολιτική, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή την υπηρεσία, καθώς και η πολιτική εμπορίου και ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία θα πρέπει να μην συμπεριληφθεί. Περιμένουμε όμως την άποψη του ύπα του εκπροσώπου και τις υποδείξεις του, γιατί εμείς δεν γνωμοδοτούμε εδώ. Νομίζω ότι η πολιτική εμπορίου και η διεύρυνση αυτής της εμβέλειας θα πρέπει να αποκλειστεί. Επίσης θα ήθελα να ε, αναφερθώ στο νομικό καθεστώς αυτής της διπλωματικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα γραφείο ή μία ε, οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει μία ε, χρηματοδοτική, μάλλον χρηματοοικονομική αυτονομία. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να είναι και οικονομικά αποδοτική. Οικονομικά αποδοτικός αυτός ο φορέας. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο θα είναι ένα ανεξάρτητο γραφείο ή ένας ε, κοινοτικός, ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο στο 5 δ στο 5D, σε σχέση με την επάνδρωση της ε, υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφανής διαδικασία, όπως ορίζει η υπεύθυνη επί του προϋπολογισμού αρχή. Αλλά επίσης, επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια, να συσταθεί μια επιτροπή επιλογής που θα ορίσει τους κανόνες έτσι ώστε να ξέρουμε ποια θεσμικά όργανα και ποια κράτη θα συμμετέχουν και πώς τα κράτη θα συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μία γεωγραφική και δημογραφική υπηρεσία και ίσως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα ίδια ε, κριτήρια αναλογικότητας που ισχύουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα πρέπει να ισχύουν και στην μελλοντική διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ότι έχουμε μία ημέρα ακόμα για την υποβολή τροπολογιών και θα την εκμεταλλευτώ. Επτά ζητούν το λόγο, επτά βουλευτές και επειδή πρέπει να τελειώσουμε στις 12.30 ε, ο καθένας σας έχει δύο λεπτά. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Σεβερίν. Ευχαριστώ. Εάν υπάρχουν κοινά συμφέροντα θα πρέπει να υπάρχει και μια κοινή πολιτική. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα και οποιαδήποτε εξωτερική πολιτική αποτελεί συγκεφαλαίωση αυτών των κοινών συμφερόντων. Το θέμα είναι ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει μια κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό που επιλέξαμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας ήταν τουλάχιστον να έχουμε μια θεσμική Υπάρχει συνοχή όταν προσπαθούμε να ε, κινηθούμε μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης. Για να είμαστε λοιπόν συνεπείς, επινοήσαμε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής, εξωτερικών υπηρεσιών που θα είναι συνεπής μόνο αν ενταχθεί τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης να υπάρχει ένας δημοσιονομικός έλεγχος επ' και την επίβλεψη του Κοινοβουλίου. Αυτή επίσης η υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξωτερικές δράσεις, δηλαδή ε, αναπτυξιακή βοήθεια, διεθνές εμπόριο και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που διαθέτει μια εξωτερική διάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση του Έλμαρ Μπρόκ, και εγώ είμαι σκιώδης για την ΑΦΚΟ, είναι πολύ καλή έκθεση. Θα πρέπει όμως να καταβάλουμε μια προσπάθεια μέχρι την τελική ψηφοφορία για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι για την κλιμακωτή εφαρμογή και την άμεση εφαρμογή την ολοκληρωτική εφαρμογή. Το θέμα δεν είναι η ουσία, το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά η έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματος, δηλαδή να γνωμοδοτήσουμε πριν απασχολήσει το θέμα το Συμβούλιο και στο τέλος θα δούμε την απόφαση του Συμβουλίου και μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Αλλά τώρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση χωρίς πολλές τροπολογίες για να κινηθούμε εντάχει έτσι ώστε το Συμβούλιο να έχει την ε, γνώμη αυτή επιτάπητος ε, όταν αρχίζει να τη συζητάει ο συνάδελφος ε, Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω τη γνωμοδότηση της κυρίας Νάιτ Σύντομα μόνο μερικές επισημάνσεις. Από τη δουλειά μου στην Επιτροπή Ανάπτυξης μπορώ να σας πω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καλύπτει και τον τομέα αυτό. Μία πολιτική έχουμε απέναντι σε τρίτες χώρες, είτε είναι αναπτυξιακή πολιτική αυτή, εμπορική ε, ή θέματα ασφαλείας. Μία είναι η πολιτική μας απέναντι στις χώρες αυτές. Γι' αυτό θα πρέπει όλα τα στοιχεία αυτά να συμπεριλαμβάνονται στην εξωτερική υπηρεσία. Στο σημείο 6 λέει σωστά η συνάδελφος ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με ζητήματα στελέχωσης και είμαι πραγματικά στεναρά πεπισμένο ότι κάθε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στέλνεται στον έξω κόσμο θα πρέπει να έρχεται προηγουμένω εδώ στην Επιτροπή μας. Γιατί όποιος μας εκπροσωπεί προς τα έξω θα πρέπει να μπορεί να αντέξει εδώ ε, τη δοκιμασία. Όποιος δίνει εδώ κακή εντύπωση ή ε, αδύναμη εντύπωση δεν μπορεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Ένα τελευταίο ε, σχετικά, ναι, όπως λέει και στο 5α, θα πρέπει να είναι ε, να υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα ήθελα να είναι και κάτι ξεχωριστό. Γιατί στον ορισμό των αντιπροσώπων να μην έχουμε την κατάσταση έτσι, ε, ε, που έχουμε ότι ε, υποβάλλονται υποψηφιότητες από διάφορες γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά τσακώνονται μεταξύ τους οι γενικές διευθύνσεις. Όχι. Και στα κράτη-μέλη δεν στέλνουμε πρέσβεις από το Υπουργείο Συγκοινωνιών ή το Υπουργείο Γεωργίας είναι διπλωμάτες οι άνθρωποι. Άρα θα πρέπει να είναι ειδικοί της εξωτερική πολιτικής. Κάπως να το ξεχωρίσουμε, γιατί να μην θεωρήσει δηλαδή το σύνολο των υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ανοίξαμε και του περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πέτσερινγκ. Κοιτάξτε, ε, εγώ μίλησα ήδη, πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης και θα καταθέσω μία τροπολογία. Πρέπει να το συζητήσω ακόμα του ε, πολιτικού μου φίλου. Ε, θα μπορούσε όμω να έχει την εξή διατύπωση. 5G, η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία οφείλει να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι συνομιλητή του στην ε, εκπροσώπησή του προ τα έξω, να διασφαλίζεται η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρένθεση, παραδείγματο χάρη οποτεδήποτε υπάρχουν διπλωματικέ επαφέ με τρίτε χώρε. Κλείνει η παρένθεση. Δηλαδή να επιμείνουμε να συμπεριληφθούμε στι δομέ ε, με σωστό τρόπο και ο κύριος Μπρόκ τα εκφράζει έτσι κάπως γενικά, αλλά θα ήταν σωστό, εν πάση κυρία συνάδελφε, να λάβετε αυτό που σας είπαμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ, κοιτάξτε, και εγώ σε γενικές γραμμές θέλω να πω ότι υπάρχει ε, συμφωνία με το σχέδιο ε, της ε, κυρίας ε, Λούνατσεκ θέλω να πω ορισμένα πράγματα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να συμπεριληφθούν. Το ένα είναι στο 5B, εκεί όπου γίνεται λόγος για το νέο θεσμικό πλαίσιο και για το, τα θέματα εκείνα που έχουν σχέση με την εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να αναφέρεται και να γίνεται αναφορά και στο περιβάλλον, την ειρήνη, την ενέργεια και εκεί υπάρχει κάποιο περιθώριο και Άρα και αυτό πρέπει να αναφερθεί. Θα σας δώσουμε την τροπολογία, απλά έτσι ήθελα να το πω ήδη τώρα. Όσον αφορά τώρα το θέμα που αναφέρθηκε σχετικά την πολιτική ανάπτυξη, να περιλαμβάνεται και αυτή στην έπειρηση. Ξέρετε ότι όλοι ασχολούνται με αναπτυξιακά θέματα. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι της αναπτυξιακής κοινότητας θεωρούν ότι δεν είναι καλό να συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη ε, γιατί θεωρούν ότι θα υποβαθμιστεί κατά κάποιον τρόπο η ανάπτυξη. Άρα δηλαδή πρέπει να συζητηθεί αυτό, κατά πόσο η συζήτηση θα είναι σωστή, η απόφαση θα είναι σωστή ή όχι. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Πέτερινγκ, δηλαδή να συμπεριληφθεί το θέμα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την ε, διπλωματική υπηρεσία, πιστεύω και αυτό είναι πολύ σωστή ιδέα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα δίκτυα υπάρχουν αυτά τα εθνικά δίκτυα και οι εθνικοί θεσμοί και όλη αυτή η διαδικασία δεν θα είναι και τόσο απλή για όσους εξακολουθούν να σκέπτονται έτσι κάπως εθνικιστικά. Η διαδικασία πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Πάντως εγώ προσωπικά τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ του να υπάρχει έτσι μια γρήγορη προσέγγιση όπως λέει και η συνάδελφος λόγω του ανταγωνισμού στον οποίο αναφερθήκατε και μια τελευταία μου παρατήρηση. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί κανείς στο ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία φύλων στην επάνδρωση της υπηρεσίας. Το λόγο έχει ε, ο κύριος Στράσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι. Κατά πρώτον όσον αφορά την ε, έκθεση ε, τη συμφωνούμε, τη στηρίζουμε και επίσης ε, ε, πράγματι ε, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μετά, πρέπει να στηρίξω αυτό που είπε ο κύριος Πέτερινγκ. Δηλαδή ότι είναι σημαντικό ευθύς εξ αρχής να καθίσταται σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εντάσσεται σε αυτό το μόρφωμα. Πρέπει αυτό να διευκρινιστεί. Το στηρίζω απόλυτα. Τρίτον, θα ήθελα να παρακαλέσω να στρέψουμε την προσοχή μας και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω ότι η έκθεση του κύριου Μπροκ προβλέπει τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Διπλωματικού Κολεγίου, ενός είδους ακαδημίας. Αυτό είναι σημαντικό ε, να υπάρχει κοινή εκπαίδευση στο μέλλον. Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες ως επ' αυτού θέλω να πω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε στη μέχρι τώρα εργασία η οποία εκφράζεται στη σταθεροποίηση ε, των δικτύων των ε, υπαρχουσών ακαδημιών. Και την εμπειρία που υπάρχει θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στην ε, στο, στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Διπλωματικό Κολέγιο ή Ακαδημία, αν θέλετε. Τελευταία παρέμβαση, πρώτη τελευταία, ο κύριος Σιμπ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νέιτς συνέταξε ένα γνωμοδοτικό έγγραφο. Έχουμε όμως και την έκθεση του κυρίου Μπροκ, κάτι το οποίο δείχνει ότι έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά ε, είναι, ε, μάλλον βρίσκονται σε μια κατάσταση διάχυσης. Θα δεχτούμε αυτό τον κατακαιρματισμό των ε, δυνατοτήτων και των πόρων μας αποφάσεις σε αυτό το τομέα πρέπει να είναι θεσμικού χαρακτήρα. Ο ε, ύπατος εκπρόσωπος θα πρέπει να συμφιλιώσει τα συμφέροντα του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το εξής και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Πέτερινγκ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενσωματωθεί στις αποστολές του Ρέλεξ, σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικών αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Βιγγένιν, ο βούλγαρος συνάδελφος, είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή γεωγραφική κατανομή Εάν δείτε τις ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του παρόντος, μπορούτε να φτάσετε σε ορισμένα συμπεράσματα ως προς τη γεωγραφική αυτή κατανομή και τη γεωγραφική διάχυση. Πιστεύω ότι αυτός ο θεσμός θα πρέπει να συσταθεί κατά τρόπο ώστε να ξέρουμε ποιος εκπροσωπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ποιος ε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελευταίο σημείο, ε, θέλω να πω κάτι σημαντικό. Υποστηρίζω αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά διαπιστώνω ότι την καταγραφή των διαφόρων σημαντικών τομέων δεν αναφέρεται πουθενά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 5β θα παρακαλούσα να συμπληρωθεί αυτό, προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι εγκάρσιο ως καθήκον ε, ε, λένε ορισμένοι και διαπερνά όλες τις ε, πολιτικές. Ναι, αλλά είναι και ανεξάρτητο και θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνεται στην εξωτερική υπηρεσία. Εγκαίρως θα υποβάλουμε και γραπτά αυτή την τροπολογία μας. Πριν ε, δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τα συμπεράσματά της, θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι την Πέμπτη η στις 12 θα πρέπει να έχετε υποβάλει τις τροπολογίες σας στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στα αγγλικά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι ευρία η συνένεση για το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τη γνωμοδότηση αυτή με την έκθεση Μπροκ για να γίνει ακόμα πιο στεναρή και ισχυρή η θέση μας. Βεβαίω, με χαρά να συμβάλλω κι εγώ στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, εάν θα καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή θέση, η προσέγγιση για το αν θα πρέπει να είναι σταδιακή η πορεία μας ή να είναι φιλόδοξο το σχέδιο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο συνολικό και φιλόδοξο φυσικά. Από εκεί και πέρα συζητάμε τις λεπτομέρειες εφόσον υπάρχει ένα γενικό σχέδιο και φιλόδοξο που μας δείχνει το δρόμο και προσδιορίζει και κάποια θέματα, τότε μπορούμε ενδεχομένως να συμφωνήσουμε για σταδιακή ε, εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Αν συμφωνήσει δηλαδή ο Έλμερ, αυτό θα μπορούσε να είναι ε, ένας ε, τρόπος να συγκεράσουμε τις διάφορες θέσεις μας. Ένα σημείο μόνο στο οποίο διαφωνώ με τον συνάδελφο Κόβατσεφ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υπηρεσία, agency ή κοινοτικό όργανο ξεχωριστό αυτή η υπηρεσία. Ε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό και θα διαφεύγει του διαρκού κοινοβουλευτικού ελέγχου, πράγμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος να μην το κάνουμε ε, υπηρεσία ή κοινοτικό όργανο. Τώρα, δημογραφική ε, ισορροπία είναι περίεργο αυτό, είναι ευαίσθητο. Ας μην μπούμε ε, στο παρόν στάδιο σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είπαμε να υπάρχει η γεωγραφική ισορροπία. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό βεβαίως. Δεν θα πρέπει να ξεχάσω επίσης και την καλή ισορροπία του φίλου uh, uh, και θα δεκτώ και αντίστοιχη τροπολογία και θα την εγκρίνω πιστεύω. Συμφωνώ με τη διατύπωση του Hans Gerd Pöttering. Όντως έχει σημασία να τονίσουμε ότι αυτές οι αντιπροσωπείες, η ε, εξωτερική αυτή υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει ε, συνδρομή και βοήθεια και στις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπήσεις και στο κοινοβούλιο. Στην αρχή νόμιζα ότι εννοούσατε να εκπροσωπείτε το κοινοβούλιο ε, στις διάφορες αυτές πρεσβείες εντός εισαγωγικών. Δεν το είχα καταλάβει καλά, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι οι αντιπροσωπείες, η εξωτερική αυτή υπηρεσία θα πρέπει να καταλάβει ότι το κοινοβούλιο είναι σημαντικό θεσμικό όργανο. Άρα είναι και στην υπηρεσία και του Κοινοβουλίου και των Ευρωβουλευτών. βεβαίω και συμφωνώ με αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα θα δούμε ότι την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως εγκάρση ας πούμε οριζόντια αρμοδιότητα ε, όπως έχει χαρακτηριστεί Ελπίζω η διατύπωσή σας να είναι ε, τέτοια ώστε να μπορέσουμε να τη δεχτούμε και να το εγκρίνουμε. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά και για την υπομονή σας κυρίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη αυτή δέσμευση που αναλάβατε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε ραντεβού στις 3 και την ψηφοφορία βεβαίως για τις, ε, τους υποψηφίους για το βραβείο Ζαχάροφ. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Χαίρετε.